Πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Παρότι πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται ακόμα σε φάση άφηξης. Όπως βλέπετε, σήμερα και αύριο νομίζω θα προεδρεύω αντί του συναδελφού Σατόρη που όπως όλοι γνωρίζουμε είχε ε, ένα θάνατο στην οικογένεια. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριξη της ημερήσιας διάταξης, την γνωρίζετε. Σύντομες ανακοινώσεις. Πρώτον, αύριο το απόγευμα η συνεδρίασή μας ε, ακυρώθηκε. Οι εργασίες μας θα τελειώσουν αύριο το πρωί, πριν το μεσημέρι. Να σας πω επίσης, όπως είδατε και πνημερίσια διάταξη, το επαναλαμβάνω, οι εργασίες μας σήμερα θα γίνουν σε αυτή την αίθουσα. Το απόγευμα και αύριο θα πάμε στην αίθουσα Γιάν 2Q2. Είδατε επίσης, σας ενημερώνω πάντως, ότι θα έχουμε σήμερα μια, το απόγευμα μια σύντομη συζήτηση, τελευταίο σημείο, για την διαδικασία ρύθμισης με έλεγχο του κανονισμού για τον καθορισμό των όγκων ε, ποσοστώσεων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου για την περίοδο 2013-2020. Σήμερα θα συζητήσουμε αυτό και αν χρειαστεί θα ψηφίσουμε. Επιπλέον να σας θυμίσω ότι θα έχουμε μια έκτακτη σύνοδο της Επιτροπής στη δεύτερη συνεδρίαση του, στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου, στις 24 Φεβρουαρίου από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ για να ψηφίσουμε ένα, το σημαντικό, σημαντικό φάκελο, το πακέτο τηλεπικοινωνιών με εισηγήτρια την κυρία Δεκαστήγιο. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Να σας πω ότι η Επιτροπή μας έχει δύο νέα μέλη. Δεν ξέρω αν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν. Ε, μία είναι παρούσα. Η κυρία Βέρα Φλασάροβα, που αντικαθιστά τον συνάδελφο Ρέμεκ που αποχαιρετήσαμε την περασμένη φορά. Καλώ ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Σύντομη θα είναι η περίοδο συνεργασία μα στην θητεία αυτή, πιστεύω ωστόσο ότι θα είναι κατά που φορά. Και ο συνάδελφο κ. Ζαλέσκι από το ΕΛΚ που θα έρθει, δεν είναι εδώ παρόν αυτή τη στιγμή, ο οποίος αντικαθιστά την συνάδελφο Κοράσκα Μπομπίνσκα και αυτός θα αποτελέσει κομμάτι της ομάδα Επιτροπή μα να σας ζητήσω επίσης να εγκρίνετε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις τα πρακτικά της συνεδρίασής μας 27-28 ε, Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνετε και προχωρούμε με την ημερήσια διάταξη που προβλέπει αυτή σήμερα το πρωί συναντήσεις πολύ σημαντικές. Συζήτηση με το Συμβούλιο και την Ελληνική Προεδρία πιο συγκεκριμένα. Έχουμε καταρχάς την επίσκεψη εδώ και τον ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε του Υπουργού κ. Χρυσοχοίδη. Διορθώστε αν η προφορά μου δεν είναι σωστή. Καλώς ήλθατε. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Εκπροσωπεί την ε, Προεδρία του Συμβουλίου που συναντήσαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Κύριε Υπουργέ, πριν σας δώσω το λόγο να θυμίσω εντάχει τον τρόπο οργάνωσης της συνεδρίασης. Έχουμε γύρω στα 45 λεπτά για να συζητήσουμε μαζί σας ε, το θέμα που μας ενδιαφέρει που είναι τα δίκτυα και ευρύτερα τις τηλεπικοινωνίες. 10 λεπτά μπορεί να είναι ο χρόνος της παρουσίασής σας κατόπιν συζήτηση με συναδέλφους και λίγος χρόνος ακόμα στη διάθεσή σας για να ανταπαντήσετε. Ευχαριστώ και καλώς ήλθατε ξανά στην Επιτροπή μας. Thank you very much. Κυρίες ε, και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας με μεγάλη χαρά και τιμή για να παρουσιάσω τα θέματα, την ατζέντα των θεμάτων της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της, των τηλεπικοινωνιών. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για έναν τομέα με πολύ αυξημένη βαρύτητα που διαμορφώνει ένα ζωτικό χώρο δράσης στο πεδίο άσκησης ε, ενεργού πολιτικής. Συνδυάζει την πολιτική με την τεχνολογία, την καινοτομία, την έρευνα, την ασφάλεια των πολιτών με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βέβαια την ανάπτυξη σε διάφορες εκφάνσεις. Έχουμε διαμορφώσει μια σειρά θεμάτων που αντανακλούν το τρίπτυχο νέες υπηρεσίες, ασφάλεια, καινοτομία, προσβασιμότητα σε όλους, σε όρους κόστους και δυνατοτήτων. Το τρίπτυχο αυτό με τη σειρά του διαμορφώνει τις προτεραιότητές μας, την προώθηση δηλαδή των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την περαιτέρω ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών και τέλος την ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων της δορυφορικής πλοήγησης. GNSS, Galileo κλπ. Η ατζέντα της ελληνικής προεδρίας περιλαμβάνει την πρόταση κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Αποτελεί ένα φάκελο μεγάλης σημασίας με ευθεία σχέση με την ενιαία ψηφιακή αγορά μέσα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διασυνοριακού και διατομιακού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ασφαλείς, αξιόπιστες και φιλικές προς το χρήστη διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές και ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων διοικήσεων. Πρόθεσή μας να συνεργαστούμε με όλους, να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για αυτό το φάκελο στο πρώτο μέρος της Προεδρίας μας, ώστε να έχουμε την έγκριση της πράξης μέχρι το τέλος αυτή της τρέχουσας μικρής και ιδιαίτερης κοινοβουλευτικής περίοδου λόγω των ε, εκλογών. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως πρόκειται για ένα σύνθετο και δύσκολο φάκελο κυρίως καθώς πολλά από τα ζητήματα που αγγίζει νομοθετούνται για πρώτη φορά. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να είμαστε ναι μεν φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστές ιδίως αναφορικά με το στόχο αυτού του κανονισμού αλλά και το βαθμό λεπτομέρειας και βάθους το οποίο επισέρχεται. Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως θα πρέπει να υπερημνήσουμε για τον απαραίτητο χρόνο για, τον, για την υιοθέτηση των σχετικών μέτρων τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από την αγορά. Δεδομένων των χρονικών περιορισμών έχουμε διαμορφώσει ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα για την πρόταση αυτή. Υπάρχει ένα σημαντικό αριθμός συναντήσεων με τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, τεχνικές συναντήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τους ε, δύο τριλόγους που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Στην ατζέτα της Ελληνικής Προεδρίας είναι επίση η νομοθετική πρόταση για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων. Η πρόταση αυτή θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των αντίστοιχων υπηρεσιών. Δράτουμε τις ευκαιρίες, χρησιμοποιώντας αυτό το βήμα σήμερα, να απευθύνω μια προτροπή προς όλους μας. Ας δώσουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας να ολοκληρώσουμε το φάκελο μέσα στην τρέχουσα αυτήν μικρή κοινοβουλευτική περίοδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο συμφώνησαν ήδη σε μια σημαντική αλλαγή. Στην αλλαγή της νομοθετικής υφής της πρότασης από κανονισμό σε οδηγία και περιμένουμε και από την Επιτροπή να υιοθετήσει την ίδια πρόταση. Η ανωτέρω εξέλιξη διευκολύνει την υιοθέτηση μιας κοινή θέση σε επίπεδο Συμβουλίου και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που θα συνεχιστεί οφείλει, όπως είπα, να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Θα ήθελα να συνεχίσω την παρουσίαση των θεμάτων της ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας αναφερόμενο σε ένα μεγάλο φλέγον πολιτικό ζήτημα της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών εν γέννη και της κυβερνοασφάλειας. Τα θέματα αυτά αποτελούν πρωτοσέλιδη είδηση πολλές φορές, σε καθημερινή βάση, διαμορφώνουν τη θεματολογία πολλών πολιτικών συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο, οι κυβερνοεπιθέσεις, η διαδικτυακή κατασκοπία, και όλα αυτά τα συναφή θέματα χρειάζονται την προσοχή μας. Ως εκ τούτου είναι ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής προεδρίας το ζήτημα αυτό, την πρόταση δηλαδή οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ελληνική Προεδρία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη πρόταση οδηγίας και θα εργαστεί σκληρά προκειμένου να υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή. Σαφώς διαμορφώνεται ένα πλαίσιο για εξαιρετικά κρίσιμες συζητήσεις γύρω από το θέμα και μια πρόκληση στην οποία πρέπει να είμαστε όλοι σε συνεχή και μόνιμη στενή συνεργασία. Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας θέσης σε επίπεδο Συμβουλίου η οποία θα δώσει στη συνέχεια τη δυνατότητα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στο δεύτερο μισό του 2014. Όμως θέλω να έρθω τώρα σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα τεράστιας πολιτικής, οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας για την Ευρώπη είναι το ζήτημα της πρότασης κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η Ευρώπη στον τομέα αυτόν στερείται σε πολλές περιπτώσεις ανταγωνιστικότητας και στοιχείων ανταγωνισμού ευρύτερα σε σχέση με άλλες μεγάλες δυνάμεις παγκόσμιες που ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες, που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες και τα οποία κατακλείζουν αυτή τη στιγμή τον κόσμο και καθιστούν και τη ζωή των ανθρώπων μέσα από την δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες της, μέσα από μια σειρά δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, που, της ανάπτυξης, της βιομηχανίας και τελικά της απασχόλησης που διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ λοιπόν είναι καθήκον μας η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μεγαλύτερες ταχύτητες, μεγαλύτερο ανταγωνισμό, μεγαλύτερη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές και εξάπλωση των τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών όλου του πλανήτη. Είμαστε εδώ λοιπόν για να σας ε, πούμε ως Ελληνική Προεδρία ότι η κοινή, η ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών αποτελεί υψίστη προτεραιότητά μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτω ώστε να προωθήσουμε όλες τις διαδικασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει, ώστε να οριμάσουμε, να προετοιμάσουμε και να οριμάσουμε την, μια τελική πρόταση, μιας και και το Συμβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ως κορυφαίο ζήτημα την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελληνική Προεδρία περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμά της και σκοπεύει να προωθήσει την υιοθέτηση ενός πλαισίου αρχών και τεχνικών για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων φορέων του δημοσίου με σκοπό το περιεχόμενο αυτό να καταστεί προσβάσιμο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα αναπηρίας, αδυναμίες ενώ ο κατάλογος των προτεραιοτήτων μας περιλαμβάνει και τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης όπως είναι το Galileo και το GNSS όπου θα προχωρήσουμε την έκδοση της καταξουσιοδότηση πράξης για τα ελάχιστα κοινά πρότυπα. Τέλος, θέλω να σας πω ότι από την Επιτροπή αυτή και κουβεδιάσαμε και χθε στην προηγούμενη Επιτροπή των Μεταφορών ε, θα περάσει το ζήτημα της μεγάλης, του μίζωνος, αν, της αν θέλετε, επιλογής των σιδηροδρομικών μεταφορών το σχέδιο που ονομάζεται Shift to Rail είναι ένα εξαιρετικής σημασίας θέμα και είναι εξαιρετικής σημασίας θέμα και γιατί η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα μέσα από υψηλής τεχνολογίας τρένα να οδηγήσει τα επόμενα χρόνια αυτήν την στροφή, να κάνει μια στροφή προς το σιδηρόδρομο για πάρα πολλούς λόγους και αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς και εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά ταυτόχρονα και είναι μια αξιόλογη πρόταση διότι συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί και θεσμικοί εταίροι στην Ευρώπη. Η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιστιτούτα, τα πανεπιστήμια, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δηλαδή ένα project στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι, είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν για να παράξουμε αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των ε, σιδηροδρομικών υπηρεσιών και της σιδηροδρομικής βιομηχανίας και ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο αλλά είναι και ρεαλιστικό. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει θέματα τα οποία είναι επεξεργασμένα, όρημα και είναι έτοιμα για να κάνουμε το επόμενο βήμα, να τα καταστήσουμε αποφάσεις στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα από όλους σας να ζητήσω να συμμετάσχουμε ενεργά στην επεξεργασία και στην ολοκλήρωση όλων αυτών των συζητήσεων έτσι ώστε να καταλήξουμε στο ποθούμενο αποτέλεσμα που αποτελεί και την υψίστη αν θέλετε, αρετή για την πολιτική. Και η, πολιτική, και η αρετή αυτή δεν είναι άλλη από το να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην υπηρεσία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και ευχαριστώ και για τη σαφήνεια της παρουσίασής σας και για το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε. Τώρα προχωρούμε στην συζήτηση. Το λόγο έχει η συντονίστρια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η συνάδελφο κ. Καστίγιο, που είναι και η συγγήτρια για την, ε, στην έκθεση που αναφέρεται και που είναι σημαντική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώ ήλθατε στην Επιτροπή κύριε Υπουργέ. Η ελληνική Προεδρία φτάνει σε μια στιγμή που ζούμε ειδικέ ε, περιστάσει από τι δραστηριότητε του Κοινοβουλίου και εν μέρει από το πώς επηρεάζει, επηρεάζουν οι ευρωεκλογές τα άλλα θεσμικά όργανα. Είμαστε στο τέλος μιας ε, κοινοβουλευτικής θητείας και στο μέσο περίπου της ε, ελληνικής προεδρίας θα διακοπούν οι κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και θα έχουμε εκλογέ. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα. Κάτω από τις περιστάσεις αυτές Μπορεί κάποιο να σκεφτεί απ' έξω ότι είναι μια προεδρία που δεν έκανε και πολλή δουλειά, γιατί στην πράξη η κοινοβουλευτική δραστηριότητα διακόπτεται, τελειώνει η θητεία του Κοινοβουλίου, άρα δεν θα υπάρχουν πολλά πράγματα να αντιμετωπιστούν. Στη συγκεκριμένη τόσο περίπτωση, το συμπέρασμα αυτό θα ήταν απόλυτα εσφαλμένο, διότι όπως πολύ σωστά εσείς στον τομέα σας ε, αναφέρατε, αλλά και σε άλλους ε, τομείς. Ε. Εμείς μιλάμε ευρύτερα για το ότι κάτω από την ομπρέλα ενιαία ψηφιακή αγορά υπάρχουν πολλές διαφορετικές πρωτοβουλίες. Τώρα, η ψηφιακή ενιαία αγορά σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες που έχει η Επιτροπή μας είναι καθοριστικές για να μπορέσει η ενιαία ψηφιακή αγορά να αποκτήσει, να γίνει πραγματικότητα. Εσείς κάνατε μια ανασκόπηση πολύ σωστά. Πολύ σωστή. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου ο ρόλος της ελληνικής προεδρίας θα είναι καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός, ούτως ώστε συγκεκριμένα ντοσιέ, η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση μπορούν να κλείσουν ή και για άλλα ντοσιέ που θα προχωρήσουν όταν ξεκινήσει η νέα θητεία με μια ε, ταχύτητα που θα επιτρέψει να ληφθούν οι αποφάσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άποψη αυτή λοιπόν αυτό που θα κάνει, που θα μπορούσε να κάνει η ελληνική προεδρία θα έχει αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον, την πορεία των προτάσεων αυτών που όπως είπα και εσείς τονίσατε και χαίρο ότι το, διότι το κάνατε, έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα για την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Θα κάνω μία σύντομη ανασκόπηση τονίζοντας κάποια θέματα που θεωρώ καθοριστικά. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ε, ε, ελληνικής προεδρίας. Είναι σε μια φάση διαπραγματεύσεων βρισκόμαστε σε μια φάση διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, διακόπτει ομιλήτρια, που επιτρέπει την, να κλείσει ο φάκελος. Αυτό θέλει η Προεδρία, αυτό θέλει το Συμβούλιο, αυτό θέλει η Επιτροπή. Δεύτερον, η πρόταση οδηγίας και για τον κανονισμό που έστειλε η Επιτροπή για την ε, ευρυζωνικότητα μπορούν να προχωρήσουν επίσης. Δύο αναφύ υπάρχουν. Εσείς αναφέρατε μία την οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων πληροφοριών που συνδέονται με τις κρίσιμες υποδομές που είναι αυτές που θέλουμε να υπάρξει εντονότερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Η Επιτροπή μας έχει κάποιες αρμοδιότητες αποκλειστικές σε σχέση με την πρόταση οδηγίας. Η άποψή μου είναι, όπως είπατε, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προχωρήσουμε σε τέτοιο βαθμό, ούτω ώστε όταν ξεκινήσει η νέα φοιτεία να λειτουργεί το Σεπτέμβριο, θα υπάρχει από πλευρά Συμβουλίου μία σειρά θέσεων που θα επιτρέψουν την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο. Σε αντίστοιχη κατάσταση, σε ένα προγενέστερο ακόμα στάδιο, είναι η πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Αγορά Τηλεπικοινωνιών. Δεν θα επιμείνω εδώ για την σπουδαιότητα, την εξαιρετική σπουδαιότητα που έχει η πρόταση αυτή για να προχωρήσει, όχι να ολοκληρωθεί, για να προχωρήσει με σημαντικά η ενιαία ψηφιακή αγορά έχει να κάνει με αυτό το σχέδιο που συζητά τώρα το Κοινοβούλιο. Είπατε και πολύ σωστά κύριε Υπουργέ και συμφωνώ με αυτά που είπατε, δεν θα φάω άλλο χρόνο, γιατί είναι τόσο σημαντική η πρόταση αυτή. Η πρόταση αυτή βρίσκεται σε κατάσταση αντίστοιχη με αυτή της προηγούμενης, την ασφάλεια των δικτύων ε, πληροφοριών, λίγο πιο πίσω. Αυτή τη στιγμή ε, δεν ψηφίστηκε ακόμα το σχέδιο στην Επιτροπή μας. Θα γίνει στις 24 του μηνός. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ που έχει αρμοδιότητες για ένα κομμάτι του φακέλου, την προστασία των καταναλωτών, θα ψηφίσει το σχέδιο αύριο εμείς θα ψηφίσουμε στις 24 Φεβρουαρίου. Και κατά πάσα πιθανότητα τον Απρίλιο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Από τη στιγμή εκείνη και μετά όταν θα έχει το Συμβούλιο σαφή εικόνα της θέσεως του Κοινοβουλίου θα ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινήσει το Κοινοβούλιο να ορίζει την θέση του, το Συμβούλιο ομιλήτρια, ε, σε σχέση με τις διάφορες προτάσεις που έχει ο κανονισμός. Με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το Σεπτέμβριο να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με αρκετά εξελιγμένη θέση και επαναλαμβάνω κύριε Υπουργέ έχει ε, τεράστιες επιπτώσεις για να μην καθυστερήσει η οδηγία περαιτέρω. Κλείνω κύριε Υπουργέ. Αντίθετα από αυτό που θα φαινόταν, η συμβολή της ελληνικής προεδρίας θα είναι σημαντικότερη από ό,τι θα ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν βρισκόμασταν σε αυτές τις ιδιαίτερες περιστάσεις της λήξης της κοινοβουλευτικής θητείας και της διακοπής των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων στη μέση σχεδόν της Προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ για την ε, θέση σας ε, που εκτιμώ ιδιαίτερα για συνεργασία με όλους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντελκαστήγιο. Η κυρία Τερέζα Μαρδουλέρα, συντονίστε των σοσιαλιστών, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Μας μένουν ε, κάποιοι μήνες ακόμα για συνεργασία μεταξύ μας. Σας άκουσα λοιπόν και με αυτά που είπατε συμπεραίνω ότι θα είναι ιδιαίτερα καρποφόρη η συνεργασία αυτή. Ε, πριν έρθει εκπρόσωπό μας για αυτά τα θέματα, παίρνω εγώ το λόγο από την ομάδα μου για να σας πω απλώς ότι σας άκουσα με σαφήνεια να λέτε ότι αν θέλουμε ανάπτυξη και αν θέλουμε απασχόληση, ανταγωνιστική. Ο τομέας της δικιάς σας ε, δραστηριότητας για μια ενιαία ψηφιακή αγορά είναι κάτι πολύ βασικό για να πετύχουμε την ανταγωνιστικότητα αυτή που θέλουμε. Ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός λοιπόν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αυτό και οι ευθύνες που έχετε είναι επίσης πολύ μεγάλες. Μας παρουσιάσατε ένα πρόγραμμα, το οριοθετήσατε πάρα πολύ καλά, φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό συγχρόνως. Αναφερθήκατε σε πολύ σημαντικά ζητήματα, τα ανέφερε και η συνάδελφος Δικαστήγιο πριν από λίγο. Και σίγουρα η συνάδελφος Χέρτζοκ επίση θα μπει περισσότερο στις λεπτομέρειες. Αυτό όμω που εγώ θέλω να σας πω είναι μια ερώτηση για τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Αναφερθήκατε σε πολύ σημαντικά θέματα για μας. Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση, για παράδειγμα. Η συνάδελφος Πιλάρντε Καστίγιο ήδη εξέγησε ποιες είναι οι δικές μας ανησυχίες επ' αυτού. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλά προβλήματα για να ολοκληρωθεί. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό και το είπατε και εσείς είναι η έκθεση για την μείωση του κόστους της ε, Τη ευρυζωνικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ζωτική σημασία να ολοκληρωθεί και αυτό το θέμα, για να το πω απλά, πριν τις ευρωεκλογέ. Ακόμα όμως δεν έχουμε επίσημη θέση από πλευρά του Συμβουλίου πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορείτε λοιπόν να μας επιβεβαιώσετε ότι η Προεδρία σας θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να πετύχει μια καλή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ακριβώς από τις επερχόμενες ευρωεκλογέ για την ευρυζωνικότητα. Και ένα άλλο σχόλιο, επιτρέψτε μου. Αυτό έχει να κάνει με το C4A. Τα GTI για μας ε, είναι όλη η συζήτηση που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 και αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Ένα από τα πλεονεκτήματα πέρα από τη συνεργασία που προβλέπετε το βασικό είναι το ότι έχουν ήδη κάνει διάφορες GTIs στο προηγούμενο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει να μάθουμε από τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα και ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που προσφέρει προς τη θέμενη αξία, όπως το είπατε κι εσείς, είναι η συνεργασία, ότι η βιομηχανία μαζί δουλεύει και δεν έχουμε ανταγωνισμό μέσα στην Ευρώπη, αλλά συνεργαζόμαστε για να μπορούμε να ανταγωνιστούμε καλύτερα προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και το Κοινοβούλιο έχει δουλέψει πολύ σε αυτό, να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και το άνοιγμα, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι έχουμε μάθει από την πρώτη γενιά. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλοι συμμετέχουν. Η επιτυχία των GTIs είναι πάρα πολύ βασικό. Αν το πετύχουμε είναι ένα εκπληκτικό μέσο πρόοδου που θα μας οδηγήσει σε ηγετική θέση όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Σε τομείς, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους συντονιστές ομάδων που έχουν ζητήσει το λόγο. Οπότε θα μπούμε στις παρεμβάσεις των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής. Ο κύριος Βιτόριο Πρώτη καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ. Θα είμαι σύντομος. Σε κάθε περίπτωση ο, μιλάμε για ευρωπαϊκές υποδομές που είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θα ήθελα να θυμίσω και το θέμα της κατασκευής ενός δικτύου ηλεκτροδότησης ε, στην Ευρωπαϊκού που θα βασίζεται σε τεχνολογίες συνεχούς υψηλής πίεσης, τάσεως. Ε, από την άποψη αυτή θα ήθελα να, ρωτήσω από να ζητήσω από την Προεδρία να αναλάβει την ευθύνη της χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των δικτύων αυτών που θα μπορούσε ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες αλλά θα μπορούσαν γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να το κάνουμε γρήγορα να φροντίσει να εξετάσει το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των δικτύων με υπομορφή ευρωμολόγων, Eurobonds. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, πιστεύω ωστόσο ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό ακριβώς διότι η εξασφάλιση ταχύτητας κατασκευής θα είχε και ε, εξαιρετικά υψηλό θετικό αντισυγκυριακό αποτέλεσμα. Αυτό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να συζητούμε σοβαρά για μια ενδεδειγμένη χρηματοδότηση στην κλίμακα των επενδύσεων. Ευχαριστώ. ο κύριος Χέρτζοκ, η κυρία Χέρτζοκ, που είναι και η συγγήτρια ακριβώς για το broadband. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο. Είχα πολύ σημαντικά καθήκοντα. Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη χαρά ορίζουμε και ακούμε την ελληνική προεδρία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους σας εδώ στις Βρυξέλλες που ήδη επομίστηκαν μεγάλο μέρος των ευθυνών ώστε με την Λιθουανική Προεδρία από κοινού να συνέλθουν και να προετοιμάσουν την Ελληνική Προεδρία σε σχέση με την αλλαγή σκητάλης για αυτά τα χαρτοφυλάκια οι συνάδελφοί σας εργάστηκαν καλά σε αυτό το επίπεδο και θα υπάρξει έτσι ανατροφοδότηση σε σχέση με τους Έλληνες Υπουργούς και αυτό είναι κάτι πολύ αξιοπρόσεκτο θα έλεγα από πλευράς Προεδρίας. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας κάποιους αριθμούς, κάποια στοιχεία. Φαίνεται ότι από τις διάφορες έρευνες ότι 250 δις ευρώ ετήσια θα μπορούσαν να προσθεθούν στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ αν είχαμε ήδη την ενιαία ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά. Όλοι γνωρίζουμε σε αυτό το σώμα ποια μάχη δίνουμε για τον ορίζοντα 2020 στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και αρκετά χρόνια. 250 δις επιπλέον όσον αφορά το ΑΕΠ Νομίζω ότι πραγματικά αυτό λέει πολλά και πρέπει να προωθήσουμε αυτή την υπόθεση. Δύο βήματα πρέπει να γίνουν. Η ψηφιακή αγορά και το ψηφιακό θεματολόγιο. Η συνάδελφος Πιλάντερ Καστίγιο ε, ε, με μεγάλη όθηση προωθούν, προωθεί αυτό το θέμα. Και το άλλο θέμα είναι υποδομές για την ψηφιακή αυτή δράση. Πρέπει να υπάρχει η ευρωζωνική αυτή διασύνδεση και δυνατότητα διαθέσιμη και δορυφορικά και με οπτικά, ε, οπτική, ε, οπτικά οπτικές ίνες. Θα πρέπει εδώ να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Θα ήθελα από πλευρά ε, των όσων λέγονται, δεν μπορούμε να ζούμε στην Ευρώπη όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν σύνδεση με το ε, διαδίκτυο και πληρώνουν υψηλότερα τέλη επειδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αγαθά ή υπηρεσίες που μπορούν να αναζητήσουν μέσω διαδικτύου. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν λοιπόν. Θα έλεγα όταν ε, δούμε τον κανονισμό αυτόν που με αφορά και αυτό που θα ήθελα να αναφέρω προσωπικά Υπουργέ είναι είχαμε διεξοδικές συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο αν θα έπρεπε να ακολουθηθεί κανονισμός ή οδηγία με τα προβλήματα που έχουμε. Αυτό όμως δεν είναι το σημαντικό για μένα. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι η ταχύτερη δυνατότητα από πλευράς διαδικασίας χωρίς καθυστερήσεις για να υλοποιηθεί αυτή η δράση. Για μένα είτε είναι κανονισμός είτε είναι οδηγία με βραχία, με σύντομη περίοδο εφαρμογής όμως για να τα λέμε ξεκάθαρα. Από το Κοινοβούλιο προς εμάς λοιπόν, αν τώρα πάμε σε οδηγία όπως αποφασίσαμε, που είναι αυτό το οποίο είχε ζητηθεί και από το Συμβούλιο, θα πρέπει να βρούμε την ε, ταχύτερη δυνατότητα υλοποίησης και εφαρμογής. Πρέπει να πάμε για απλούστευση, να πετύχουμε την απλούστευση. Απλουστεύοντας τα πράγματα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Περιπλέκοντάς τα δεν μπορεί να γίνει σωστά η δουλειά. Πρέπει να επιτευχθεί η πρόοδος για να έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο. Υπουργέ, εγώ προέρχομαι από την Ουγγαρία. Πριν από 10 χρόνια για μας ε, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν υπό την, ε, ε, η ευρωπαϊκή διεύρυνση που επετέφθη. Όταν ε, οι χώρες αυτές εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπόρεσαν έτσι να ευδοκιμήσουν, τις, να ευδοκιμήσουν οι προσπάθειες που είχαν γίνει. Λοιπόν, σε σχέση με την Ευρώπη, για τη διασύνδεση που θα πρέπει να επιτευχθεί και πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Έχετε μια νέα δυνατότητα νέα διεύρυνση λοιπόν από πλευρά τη Ελληνική Προεδρία. Ευχαριστώ. Ehm. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιουτικόφερ, ευχαριστώ Υπουργέ. Εγώ συμφωνώ πρέπει να πω και μάλιστα πλήρως με αυτά τα οποία η συνάδελφος από την Ουγγαρία προανέφερε για υποσχέσεις ε, για μια ολοκληρωμένη αγορά σε σχέση με τα ψηφιακά στην Ευρώπη. Θα ήθελα όμως να προσθέσω εδώ μια διαφοροποίηση, ένα ευαίσθητο ίσως πολιτικό ζήτημα, το οποίο αναφύεται σε πολλές δημόσιες συζητήσεις ε, μέσα στο πλαίσιο των ανησυχιών μας ε, για την κατασκοπία που διεξάγεται από την NSA από πλευρά των ΗΠΑ της ε, Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας και άλλους. Έγινε λόγος για ευρωπαϊκές λέει που πρέπει να υιοθετηθούν δεν θα μπορούσαμε να διευρύνουμε το πεδίο ασφάλειας της προστασίας προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, υιοθετώντα μια ευρωπαϊκή λύση κάπως, την οποία θα προσεγγίζαμε. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Και όταν φυσικά κάνουμε λόγο για μια ενιαία εσωτερική αγορά, δεν έχουμε ακόμα διευθετήσει το θέμα ποιος θα ήταν, ποιοι θα ήταν οι παίκτες που θα εμπλεκόντουσαν σε αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά. Ποιοι θα έδρεπαν τους καρπούς και θα υποφελούντο θα έχουμε Ευρωπαίους παίκτες που θα ήταν ακόμα και σχεδόν στο ύψος των περιστάσεων για να παρέχονται αποτελεσματικές ε, λύσεις ε, και υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που θα ε, λάμβαναν υπόψη περισσότερο τα θέματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων από ό,τι σε σχέση με άλλους κατά το παρελθόν. Το ερώτημα προς εμάς λοιπόν Υπουργέ είναι και αυτό γνωρίζω ότι είναι πολιτικού χαρακτήρα ερώτημα, είναι υπάρχουν κάποιες υποσχέσεις καθότι εσείς μπορείτε να δείτε σε αυτή την προσέγγιση υποσχέσεις που θα μπορούσαν να δοθούν. Δεν θέλω να, ακούσω, να ακουστώ επιφυλακτικός ε, και σκεπτικιστής, αλλά για μια προσέγγιση ευρωπαϊκού χαρακτήρα υπάρχει κάποια προσδοκία, κάποια υπόσχεση προσδοκία σας σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς βλέπετε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έκλεισαν ο κύκλο των παρεμβάσεων. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό για να ανταπαντήσει. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Πολύ ε, όλους και όλες για την ε, συμμετοχή σας στην ε, συζήτηση αυτή. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αντελκαστίγιο η οποία με πολύ προθυμία και με πολύ μεγάλη προσπάθεια επιχειρεί να συντάξει μια πρόταση μέσα από τη δημιουργία ε, των αναγκαίων ισορροπιών έτσι ώστε να καταλήξει σε μια πρόταση κοινά αποδεκτή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί της έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε δύο μήνες, τώρα βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε, σε δύο μήνες πρέπει να κάνουμε πράγματα που οι άλλες προεδρίες θα κάνουν σε έξι μήνες διότι η δική μας Προεδρία έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα των εκλογών. Για το θέμα της ε, κοινή αγοράς τηλεπικοινωνιών θα αρχίσουμε να εξετάζουμε ενδελεχώς την πρόταση στο Συμβούλιο ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια υψηλή πολιτική ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το κόστος τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών δικτύων και το κόστος ανάπτυξης των ε, δικτύων έχει αρχίσει ήδη εντατικά η εξέταση από το Συμβούλιο και στις 30 Ιανουαρίου η Προεδρία θα ζητήσει εντολή διαπραγματεύσεων από το Κορεπέρ ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί οι τρίλογοι και οι τεχνικές συναντήσεις. Συνεπώς θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε, θα πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά την ε, ερώτηση της κυρίας Χέρτοκ από την Ουγγαρία, η συναδέλφου. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Προσπαθούμε εντατικά για την επίτευξη των στόχων όλου του ψηφιακού θεματολογίου. Η μείωση του κόστους των δικτύων, της ανάπτυξης των δικτύων είναι η δεύτερη προτεραιότητα και συμφωνούμε απόλυτα στην υιοθέτηση της πρότασης. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και φυσικά θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση για το χρόνο εφαρμογής μεταφοράς στα εθνικά δίκαια. Ε, βέβαια, εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και ένα πολιτικό θέμα διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το shift to rail, πραγματικά το shift to rail, το θέμα αυτό, δίνει τη δυνατότητα στη βιομηχανία και στην έρευνα να εργαστούν μαζί αρμονικά και να παράγουν αποτελέσματα. Σήμερα γίνεται η παρουσίαση του προγράμματος στη σχετική ομάδα εργασίας από την Προεδρία μας. Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε όλοι μαζί έχοντας την εμπειρία και τη γνώση από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και να δημιουργήσουμε μια σημαντική δομή για το σιδηροδρομικό τομέα. Είναι άλλωστε, όπως είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, στην πρώτη μου ομιλία, βασική πολιτική επιλογή για τις μεταφορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Μπουτικόφερ σχετικά με την ε, με, την, ε, το μεγάλο ζήτημα της προστασίας των δεδομένων, της ασφάλειας των επικοινωνιών, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε τα τον τελευταίο καιρό ε, αναφέρθηκα στην αρχή στον τρόπο με τον οποίο η Προεδρία θα προσπαθήσει το επόμενο διάστημα να προχωρήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες για την πρόταση για αυτό που ονομάζεται κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια τηλεπικοινωνιών. Ε, έχω θητεύσει ε, πολλά χρόνια υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας στη χώρα μου. Και θέλω να σας πω από την εμπειρία που διαθέτω χρειάζονται τρία πράγματα για να γίνουμε απολύτως πρακτικοί και όπως είπα να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες αλλά να γίνουμε χρήσιμοι και για την ασφάλεια των χωρών μας, την ασφάλεια της Ευρώπης και τη θωράκιση. Το πρώτο που χρειάζεται είναι κανόνες, οι οποίοι κανόνες θα έχουν, έχουν να κάνουν με το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και την, και την εθνική ασφάλεια που αφορά κάθε χώρα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την διαρκή επαγρύπνηση που πρέπει να διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μηχανισμούς της ούτως ώστε κάθε φορά επειδή αναπτύσσονται οι τεχνολογίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολλές φορές η ανάπτυξη των τεχνολογιών και η αύξηση των προβλημάτων γίνεται πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατή επίλυση και αντιμετώπιση τους. Χρειάζεται λοιπόν μια, ένας μηχανισμός διαρκούς επαγρύπνησης, αναθεώρησης και τελικά το τρίτο που χρειάζεται και το πιο σημαντικό για μένα, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτούνται καθημερινοί ...θεσμοθετημένη έλεγχη. Αυτό το οποίο λείπει από τα ζητήματα αυτά είναι ο έλεγχος. Διότι πολλές φορές η έλλειψη ελέγχου, η έλλειψη ή μάλλον η αδράνεια που διακρίνει τους μηχανισμούς οδηγεί σε τεράστια προβλήματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα κάτω από τα πόδια μας ή αυτά που περνάνε μπροστά μας, σαν το, ποτάμι, το νερό από το ποτάμι, έχουμε, είμαστε παρατηρητές και δεν βλέπουμε ότι ακριβώς εκείνη την ώρα αναπτύσσονται προβλήματα τα οποία έπρεπε ήδη να είχαμε αντιμετωπίσει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε, έχουμε βάλει ως προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, σε ό,τι αφορά την, ε, αυτό που λέγεται κυβερνοασφάλεια, να καταλήξουμε τον Ιούνιο είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ξέρετε ότι χρονίζει. Θα κάνουμε το, το θέμα του data protection δηλαδή. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τουλάχιστον από την Ελλάδα έχουμε στείλει τους καλύτερους εμπειρογνώμονες για να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Όμως κάνω μια έκκληση ότι όλες οι χώρες όχι μένω μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη επιτροπή αλλά και τις επιτροπές όλες εκείνες και τα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με την ασφάλεια και τη θωράκιση της ε, συνολικότερης ασφάλειας της Ευρώπης να είναι άγρυπνοι και να παρακολουθούν αφενός με τις εξελίξεις τις τεχνολογικές και από την άλλη οι μηχανισμοί του ελέγχου να είναι διαρκώς επαγρύπνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή συζήτηση. Καλή δύναμη. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και την ομάδα σας βεβαίως. Ε, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίσατε και εκθέσατε αυτά το πολύ σημαντικ, τους πολύ σημαντικούς φακέλους. Όπως καταλάβατε η Επιτροπή μας θα σας δείξει ότι όσο μεγαλύτερη συνεργασία γίνεται ευχαριστούμε εκ νέου.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 Allora c'è un piccolo capannello. Bene, e diamo... Ωραία. Καλωσορίζουμε εκ νέου την ελληνική προεδρία, αυτή τη φορά στο πρόσωπο του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, Υπουργού Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα και θεμάτων δηλαδή που βρίσκονται στο κέντρο των εργασιών τη Επιτροπή μα και των γενικότερων συμφερόντων της Ένωσης. Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω το λόγο. Σας καλωσορίζω. Είμαι βέβαιο ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά μαζί. Παρότι έχουμε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα σε αυτή την ιδιαίτερη θεσμική στιγμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που όπως ξέρετε αποτελούν, οι εκλογές αποτελούν κεντρικό σημείο του εξαμήνου. Θα σας ε, δώσω το λόγο για να κάνετε μια παρέμβαση, κατόπιν οι συνάδελφοι υποβάλλουν ερωτήματα παρεμβάσεις και εν τέλει θα έχετε ξανά το λόγο για τελικά σχόλια. Παρακαλώ. Thank you, President. President. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Ήτρε, αγαπητοί φίλοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Και αυτό γιατί ήμουν εγώ ο ίδιος ευρωβουλευτής για 13 χρόνια. 1994 με 2007. Συνεπώς, μέρος της καρδιάς μου εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ, μαζί σας. Και δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα για το Συμβούλιο. Να είναι προεδρεύων του Συμβουλίου Ανταγωνισμού κάποιος που έχει περάσει τόσα χρόνια εδώ, μια που υπάρχει κάποιο είδου ανταγωνισμό ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δεν ξέρω τελικά αν εξυπηρετώ τα συμφέροντα δηλαδή του Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου. Τέλο πάντων, αστείευομαι όπω καταλαβαίνετε. Τη Ευρώπη. Σωστό, σωστό. Τη Ευρώπη τα συμφέροντα στηρίζω. Εν πάση περιπτώσει, όπω γνωρίζετε, η Ελληνική Προεδρία είναι μια ιδιαίτερη Προεδρία. Αυτή συγκεκριμένη, γιατί όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία ουσιαστικά κρατάει τρεις μήνες μόνο, εξαιτία των ευρωεκλογών ακριβώς. Δεν έχουμε λοιπόν ψευδεστήσεις. Γνωρίζουμε ότι είναι μια ιδιαίτερα φορτωμένη προεδρία. Γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα. Και τρίτον, γνωρίζουμε ότι προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να επικεντρωθούμε στα διάφορα ζητήματα και να έχουμε απτά αποτελέσματα. Αυτή είναι και πρόθεση του Πρωθυπουργού και ολόκληρη τη ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να είναι μια προεδρία που έχει σαν στόχο αποτελέσματα. Πράγματι, ο στόχος μας, για να το πω με άλλα λόγια, είναι να εκπλήξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και όλους τους μετέρους με θετικό τρόπο. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πραγματιστές και όντως να αποδώσουμε με αποτελέσματα. Φυσικά η βιομηχανική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα κλειδί για την ελληνική προεδρία. Το ίδιο ισχύει και για το Συμβούλιο ολόκληρο βέβαια και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό συμβαίνει γιατί η βιομηχανική πολιτική αποτελεί ένα εργαλείο κλειδί για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας και να ξεπεράσουμε την τρέχουσα κρίση. Παρόλο που η βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί την ε, δραστηριότητα η οποία βοηθάει με 34 εκατομμύρια θέσει απασχόληση έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την κρίση και αντιμετωπίζει προκλήσεις ανταγωνισμού από αναδυόμενες αγορές. Το τμήμα του ΕΠ έχει πέσει από τα 15,5% που ήταν το 2012 σε 15,1% το 2013, ενώ ο στόχος είναι 20% για το 2020. Συγχρόνως έχουμε 3,8 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν από το 2008 μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει και να ενισχύσει την θέση της στον κόσμο. Περιτώ να πούμε ότι η ελληνική βιομηχανία αποτελεί θύμα της κρίσης αυτής. έχουμε ειδίκευση σε θέματα μεταποίηση τροφίμων, επεξεργασία τροφίμων μάλλον, ε, φαρμακευτικών, μετάλλου, χημικών, τσιμέντου και φαντουργίας. Όμω τα τελευταία έξι χρόνια η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 35% και τώρα αποτελεί μόνο το 9% του ελληνικού ΑΕΠ, πολύ πιο χαμηλά δηλαδή από τα 15,5% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μεγάλοι τομείς, όπως ο οικοδομικός τομέας και οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν πολύ ενέργεια, έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ σοβαρά και από την μείωση της ζήτησης, αλλά και από τις υψηλές τιμές στην ενέργεια. Τώρα, θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, συμβολή της βιομηχανίας στο Ευρωπαϊκό ΕΠ κατά 20%. Στόχος όμως που δεν είναι εύκολος, ούτε προφανής. Και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της ε, ετήσιας έρευνας, ε, έκθεσης μάλλον για τον ανταγωνισμό. Η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται, οι περιφερειακές ανισορροπίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Η κοινωνική συνοχή επίσης υποφέρει πολύ εξαιτία της συνεχιζόμενης ύφεση και τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ανευπρεγουμένου στην ανεργία. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι προφανές. Επίγει να βάλουμε πάνω πάνω στην ημερήσια διάταξη μια ανανεωμένη βιομηχανική πολιτική τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το έχουμε συζητήσει άτυπα αυτό με άλλους υπουργούς και πρέπει να ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το θέμα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα και θα συζητηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον επόμενο Μάρτιο και στα πλαίσια επίσης δύο Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας του επίσημου το Φεβρουάριο εδώ στις Βρυξέλλες και του άτυπου που θα λάβει χώρα στην Αθήνα το Μάιο. Το μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη του άτυπου Συμβουλίου αυτού του Μαΐου θα είναι η βιομηχανική πολιτική. Το λέω αυτό για να υπογραμμίσω πόσο μεγάλη σημασία έχει το θέμα αυτό σε σχέση με τον τελικό μας στόχο που είναι νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις απασχόλησης, κυρίως βέβαια για τους άνεργους. Οι συζητήσεις εννοείται ότι θα βασίζονται στην ανακοίνωση που θα υιοθετηθεί σήμερα, κατά σύμπτωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική και θα λαμβάνει υπόψη και τις διάφορες ανακοινώσεις που έχουν γίνει για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Θα βασίζεται επίσης και στο RISE, την ε, έκθεση που πρόσφατα υιοθετήθηκε. Έχουμε εδώ τον εισηγητή, τον κύριο Μπετικόφερ. Η Ελληνική Προεδρία καλωσορίζει την έκθεση αυτή, RISE, η οποία αναφέρεται σε θέματα τεχνολογικά, περιβαλλοντικά, ε, κοινωνικής κοινοτομίας και μας οδηγεί στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση μέσω μιας αποτελεσματικής στρατηγικής που επαναβιομηχανοποιεί την Ευρώπη, ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία συνολικά και αντιδρά με υπεύθυνο τρόπο στις νέες κοινωνικές προκλήσεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι οι κατασκευέ είναι ένας τομέας ο οποίο αναγνωρίζεται ότι αποτελεί την κινητήρια δύναμη της σύγχρονης οικονομίας. Συνεισφέρει πολύ στην παραγωγικότητα, συνεισφέρει στην έρευνα, στην καινοτομία, που είναι τέσσερις φορές παραπάνω σε σχέση με το ΕΠ και έχει και πολλαπλαστικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη και στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. Συνεπώς, αν πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό σημαίνει ότι θα μεταρρυθμιστεί το βιομηχανικό μοντέλο, τονίζοντας ιδιαίτερα την κοινοτομία, την καινοτομία και την ε, διεθνοποίηση. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όσον αφορά τον πιο νέο παραγωγικό πληθυσμό που πλήττεται τόσο πολύ από την κρίση θα βοηθηθεί διότι θα έχουμε νέα παιδεία που μπορούν να προσφέρουν ενέστες απασχόλησης. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία ακόμα και σε πιο παραδοσιακούς τομείς και τρίτον θα αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας με προσανατολισμό τις εξαγωγές. Και εδώ θέλω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Η Προεδρία θα επικεντρωθεί σε πέντε αρχές κυρίως. Η πρώτη αρχή είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση του επιχειρησιακού κλίματος. Πρέπει να τροποποιήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει να μειώσουμε το άχθος που πέφτει στους ώμους των επιχειρήσεων και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Εντοπίζοντας λοιπόν τέτοια νομοθεσία θα απλοποιήσουμε και τις διαδικασίες και θα έχουμε ένα πιο σταθερό φορολογικό σύστημα, κάτι το οποίο θα συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στους στόχους μας. Αυτό είναι ο πρώτος μας στόχος. Δεύτερον, θέλουμε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του υψηλού κόστους ενέργειας. Είναι στοιχείο κλειδί αυτό κατά τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει δυστυχώ μια ενωπημένη ενεργειακή αγορά, κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αν προωθήσουμε λοιπόν μια τέτοια αγορά, αυτό ήδη είναι αναγκαίο και σίγουρα θα βοηθήσει πολύ. Έπειτα, πρόσβαση σε οικονομικά μέσα. Να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την βιομηχανία που πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Πρέπει να είναι ευέλικτο το μέσο αυτό, ώστε στο τέλος να μπορούν εύκολα να το χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Δεν χρειαζόμαστε δηλαδή ένα νέο γραφειοκρατικό μέσο, χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά στι ανάγκε τη αγορά. Πρέπει δηλαδή να είναι προσανατολισμένο στι ανάγκε τη αγορά. Τέταρτον, θέλουμε να δώσουμε όθηση στι επενδύσει στην καινοτομία. Καινοτομία είναι η λέξη κλειδί. Και αυτό σε συνδυασμό με την ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο έχει συζητήσει τον Οκτώβριο που μας πέρασε το Συμβούλιο, από ό,τι θα θυμόσαστε. Πρέπει η Ευρώπη να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την ικανότητά της για καινοτομία και να την απορροφήσει επίσης. Πέμπτη προτεραιότητά μας είναι η ανάπτυξη δεξιοτεχνιών, προσόντων, που χρειάζονται σε αναδυόμενους βιομηχανικούς τομείς και αγορές. Πρέπει να επενδύσουμε σε μια οικονομία της γνώσης Συνεπώς οι δεξιοτεχνίες είναι αναγκαίες για να εντοπιστούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Πετυχαίνοντας όλους αυτούς τους στόχους, εξορισμού πιστεύουμε, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εννοείται ότι δεν είναι εύκολο. Εννοείται ότι δεν πρόκειται για κάτι που θα γίνει έτσι αυτόματα. Θα χρειαστεί και χρόνος και θάρρος. Πρέπει όμως να δράσουμε και να δράσουμε τώρα. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα γιατί αντιμετωπίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα της σημερινής ευρωπαϊκής βιομηχανίας αντιμετωπίζουμε και το θέμα της ανεργίας. Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μια κοινωνική πολιτική ουσιαστικά τελικά. Τέλος, είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κοιτάμε την βιομηχανική πολιτική σαν μια συνολική προσέγγιση. Δεν πρέπει δηλαδή να βάζουμε όρια, σύνορα μεταξύ επιτροπών, γενικών διευθύνσεων, συμβούλων κλπ. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο συνεκτική προσέγγιση σε σχέση με τη βιομηχανική πολιτική και τις υπόλοιπες πολιτικές, είτε αυτή είναι η ενεργειακή, είτε είναι η περιβαλλοντική, είτε είναι της έρευνας, της καινοτομίας, του εμπορίου, του ανταγωνισμού και της εσωτερικής αγοράς. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε επιγόντως για να έχουμε στα χέρια μας μια προστιθέμενη αξία για τις πολιτικές μας. Η κατακαιρματισμένη προσέγγιση δεν βοηθάει καθόλου. Αντίθετα. Συνεπώς, για να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι είναι σαφές πως η βιομηχανική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα κλειδί, όχι μόνο για το Συμβούλιο Ανταγωνισμού, αλλά γενικά για την ελληνική Προεδρία, στο σύνολό της. Έχουμε δύο συμβούλια ανταγωνισμού αφιερωμένα στην πολιτική αυτή και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Αυτό είναι το πρώτο μου συμπέρασμα. Δεύτερο, πρέπει να δράσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εννοείται, γι' αυτό και η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά επίσης και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος, οι συντονιστές, οι εισηγητές τα μέλη της Επιτροπής. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε μαζί, να εξετάσουμε τις απόψεις σας, να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις σας. Γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό το θέμα. Τρίτο, τρίτη παρατήρηση είναι ότι δεν υπάρχουν θαύματα στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή και μάλιστα όχι σε τρεις μήνες, πόσο μάλλον, ή έστω σε έξι μήνες. Όμως, θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και συστηματικά, προκειμένου να έχουμε ορατή πρόοδο. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Δεν πιστεύουμε ότι πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα μέχρι τον Ιούνιο. Καθ' άλλο. Όμως θέλουμε μια επικοδομητική προσέγγιση, θέλουμε να δράσουμε καταλήτικα ώστε να πετύχουμε κάποια πρόοδο, ώστε να φτιάξουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτός είναι και ο στόχος μας, να έχουμε πρόοδο μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ώστε η Ιταλική Προεδρία που θα ακολουθήσει, η Νέα Επιτροπή και το Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουν να υιοθετήσουν νέα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν θέματα κλειδί που έχουν να κάνουν με την βιομηχανική πολιτική. Συνεπώς, η βιομηχανική πολιτική είναι προτεραιότητα κλειδί για μας. Θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με εσάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή Ήτρε. Και δεν έχουμε... Πιο πολύ μάλλον επικεντρωνόμαστε στο ρεαλισμό προκειμένου να κάνουμε κάποια βήματα μέχρι τα τέλη του Ιουνίου και δεν λέμε ότι θα τα καταφέρουμε όλα. Και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά είναι το ότι στηρίζοντας τη βιομηχανία δεν κάνουμε καλό μόνο στη βιομηχανία. Κάνουμε καλό σε ολόκληρη την κοινωνία, σε ολόκληρη την οικονομία και ιδιαίτερα σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Γι' αυτό η βιομηχανική πολιτική αποτελεί προτεραιότητα κλειδί για την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ε, εξαιρετικά διαφωτιστική παρουσίασή σας. Είμαι βέβαιη ότι η προηγούμενη εμπειρία σας ε, στο Κοινοβούλιο θα σας βοηθήσει, δεν θα σας εμποδίζει για να έχουμε μια ουσιαστική συνεργασία. Αντί των συντονιστών που δεν είναι παρόντες, διακόπτει η ομιλήτρια, θα δώσω το λόγο εξ ονόματος των ομάδων. Ξεκινούμε με την ε, κυρία, με τους διάφορους εισηγητές. κυρία Τζόνταν. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε και πάλι Υπουργέ κύριε Χατζηδάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ απόλυτα με τις προτεραιότητες σας, τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Είπατε ότι θα έχετε μόνο τρεις μήνες νομοθετικού έργου στην Προεδρία σας ως χρόνο, από πλευράς χρόνου. Θα είναι όμως πολύ σημαντική αυτή η περίοδος, διότι υπάρχουν πολιτικές που δεν είναι οδηγίες ή νομοθετικά έγγραφα, αλλά οι συζητήσεις για αυτά τα έγγραφα, οι συζητήσεις αυτές μπορούμε να καθορίσουμε ακόμα τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο. Το πρόβλημα ή πρόκληση για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα είναι ότι εξαρτάται από πολλές άλλες ε, πολιτικές και στοιχεία, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, την ενέργεια, κλιματικά, κλιματολογικά θέματα, εσωτερικής αγοράς κτλ. κτλ. Για μας ε, ως ε, ομάδα, κοινοβουλευτική ομάδα, το θέμα της ανταγωνιστικότητας ήταν πάντα και είναι πάντα τεράστιας σπουδαιότητας όπως είπατε δεν είναι μόνο το κέρδος της οικονομίας από αυτές τις δράσεις, αλλά είναι η βάση, τα θεμέλια για νέες θέσεις απασχόλησης, για την ευημερία, κοινωνική ευημερία, περιβαλλοντικά, για περιβαλλοντικά θέματα κτλ. Όλα τα σύναφη. Θέλω να υπογραμμίσω την σπουδαιότητα του πακέτου ενέργειας για το 2020 ως χρονοορίζοντα. Θα έχετε στοιχεία και σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά Έχουμε συζητήσει και με τους άλλους συναδέλφους σας υπουργούς επ' αυτού του πεδίου. Όμως αυτό, μια και έχει τέτοια τεράστια επιρροή και με τέτοια εμβέλεια και για την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανία. Θέλω να σας ζητήσω να μας πείτε για το όραμά σας. Πώς εσείς βλέπετε αυτή την πολιτική, κλιματολογικές αλλαγές, ενεργειακή πολιτική, μέχρι έναν ευρύτερο χρονορίζοντα. Πώς το βλέπετε εσείς στο πολιτικό επίπεδο, το έργο που ακολουθείτε για να ολοκληρωθεί η αηφόρος ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να, επιτευχθεί, ε, να επιτευχθούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και παρόλα αυτά να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε υψηλή υψηλή ανταγωνιστικότητα για τις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε τις ενεργειακές τιμές, τιμές ενεργειακών προϊόντων. Επισκέφθηκα κάποια από τα μεγάλα, κάποιες από τις μεγάλες ε, βιομηχανίες ε, στην Ευρώπη και μου είπαν ότι οι ενεργειακές τιμές είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά τους. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα ποιες συγκεκριμένες εξειδικευμένες δράσεις προγραμματίζετε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αναφέρατε το, τον τομέα των ε, συναφών θεμάτων όσον αφορά τα θέματα διαρροής ε, άνθρακα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, μια και αφορά την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το όραμά σας αυτό το θέμα. Και ένα τελευταίο θέμα. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε μια έκθεση για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Ο κύριος Μπιουτικόφερ ήταν εισηγητής για αυτήν την έκθεση. Είμαι βέβαια ότι θα αναφερθεί το θέμα αυτής της έκθεσης πολύ σχηδός. Θα ήθελα να ακούσω όμως ποια είναι η δική σας αμφίδρομη δράση επ' αυτής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές, ο συνάδελφος κ. Λάγκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος εδώ σε αυτή την αίθουσα που να είχε κάποια ένσταση ή αντίρρηση για τα όσα μας εκθέσατε. Όμως ωστόσο είναι σημεία όλα αυτά τα οποία δεν είναι καινοτόμα, δεν είναι καινούρια. Ήδη είχαμε την πρώτη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010 που μας υπευλήθη και μετά συνέταξε έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, ήμουν εγώ εισηγητής το 2011, είχαμε μια δεύτερη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακολούθησε, μετά ο Beauty Coffee συνέταξε έκθεση και τώρα έχουμε σήμερα την τρίτη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν τα δει κανείς όλα αυτά από κοινού, διαπιστώνει κανείς ότι ουσιαστικά Πολλά ωραία λόγια διατυπώνονται και διακηρύσσονται, αλλά δεν ακολουθούν συγκεκριμένες δράσεις, χειροπιαστά μέτρα. Και ο Γερμανός ποιητής Γκέτε είχε γράψει ήδη στο παρελθόν ότι αρκετά λόγια ακούσαμε. Τώρα αυτό που πρέπει να δούμε είναι πράξεις. Και διαρωτώ Ποια είναι τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα μέτρα ώστε η βιομηχανία να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί. Ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα ώστε το πολιτικό, τον πολιτικό στόχο το 2020 πραγματικά να έχουμε 20% που θα αφορά το βιομηχανικό μας προϊόν. Και βλέπω ελάχιστα πράγματα δυστυχώς να πάρει ευχή πρέπει να το πω ελάχιστα πράγματα και χρειάζονται κάποιες ενδείξεις. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα καταφέρουμε. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω εμείς να έχουμε για παράδειγμα έναν έλεγχο για την ανταγωνιστικότητα, βιομηχανική ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη που να είναι δεσμευτικός αυτός ο έλεγχος, με δεσμευτικούς δείκτες. Ούτε βλέπω το μέσο του άρθρου 170 να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη ως προς ανατολισμοί που στη συνέχεια τις δικές σας ε, βιομηχανικές πολιτικές θα τις οδηγούν σε μια μεγαλύτερη σύγκληση. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη ανακοίνωσή της τουλάχιστον το είχε σκιαγραφίσει ότι θα γινόταν και ένα ε, συμβούλιο για θέματα ανταγωνισμού είχε θυγεί αυτό αλλά μέσα σε τέσσερα χρόνια από τότε, τότε δεν ακολούθησαν κατευθυντήρες γραμμές ως προς ανατολισμοί για τα κράτη-μέλη και πώς μπορεί να ακολουθήσει κανείς μια λογική αποτελεσματική πολιτική για τον ανταγωνισμό όταν πολλά ωραία λόγια ακούγονται αλλά όμως τα κράτη-μέλη στη συνέχεια δεν καταλήγουν σε μια κοινή προσέγγιση για την ενίσχυση της βιομηχανικής τους πολιτικής από κοινού. Δεν υπάρχει σύγκληση. Γι' αυτό έχω πραγματικά έντονο αίτημα, παράκληση. Όχι να ακούμε και να χάνουμε τα λόγια μας σε ωραίες διατυπώσεις, σε πολλά λόγια, αλλά συγκεκριμένα εξειδικευμένα μέτρα να υποβληθούν ως προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπουτικόφ για ε, πράσινους, ε, τον έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Χατζηδάκη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιστρέψατε σε αυτό και καλώς ορίσατε πάλι κύριε Υπουργέ. Για τα όσα είπατε, για την στεναρή δέσμευσή σας ε, για την βιομηχανική πολιτική χάρηκα φυσικά και φυσικά για τα, ε, τα καλά λόγια για την έκθεση που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο και για την προσφορά σας για συνεργασία μαζί μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πρέπει όμως από την άλλη πλευρά ωστόσο να εκφράσω και την απογοήτευσή μου. Να την εκφράσω την απογοήτευσή μου για τον εξής λόγο. Επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν κάνω λόγο για, το, την δουλειά της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο, κάνω λόγο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμεινο μια αρχικά με μεγάλη προϊστορία και πολλές τυμπανοκρουσίες ε, βιομηχανική σύνοδο την ακύρωσε. Και τώρα φυσικά το Φεβρουάριο θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη βιομηχανική πολιτική, σίγουρα. Φοβούμαι όμως, αν διαβάζω καλά και ερμηνεύω σωστά τα μηνύματα, ότι η βιομηχανική πολιτική τον Φεβρουάριο θα συρρυκνωθεί. Θα συρρυκνωθεί σε δύο θέματα το πολύ πολύ. Ενεργειακές τιμές και απορρίθμιση και άκουσα πολύ προσεκτικά τι είπατε, ότι το δικό σας θεματολόγιο δεν συρρυκνώνεται σε μόνο αυτά τα δύο θέματα, αλλά έχετε ένα πεδίο, ένα φάσμα ε, θεματολογίου ευρύτερο και το βρίσκω αυτό πολύ σωστό και δίκαιο. Μόνο πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε από την άλλη πλευρά ότι στη βιομηχανική πολιτική, και εδώ προσθέτω τη φωνή μου στα όσα είπε ο συνάδελφος Λάγκε, δεν θα έχουμε μόνο διακηρύξεις και δεκάρικους κυριακάτικους λόγους σε κηρύγματα, αλλά θα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα και χειροπιαστά πράγματα για το Συμβούλιο Ανταγωνισμού. Ξέρετε ότι ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη και κάποιοι Υπουργοί Οικονομικών στα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια υπέβαλαν προτάσεις. Πώς μπορεί κανείς το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας να το ενδυναμώσει και να το ενισχύσει σίγουρα λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα οποία εσείς ο ίδιος αναφέρατε ότι εδώ πρόκειται για ένα εγκάρσιο οριζόντιο συνολικό τέτοιο εγχείρημα και όχι κατακαιρματισμένο μπορείτε εσείς λοιπόν στο χρόνο της ελληνικής προεδρίας να υποβάλλετε συγκεκριμένες χειροπιαστές προτάσεις για τη διακυβέρνηση governance για να υπάρξουν μέσα ώστε οι πολλές καλές ιδέες που βρίσκονται μετέωρες και εκκρεμούν να μπορέσουν να προσγειωθούν και να λειτουργήσουν και να μην βρίσκονται ε, εθεροβάμονες ε, ε, μετέωρες. Και όσον αφορά τις προτεραιότητες που μας αναφέρατε, κάποιες από αυτές τις προτεραιότητες σίγουρα θα είναι προτεραιότητες όταν εσείς δεν θα είσαστε πλέον υπουργό και όταν εγώ δεν θα είμαι πλέον ευρωβουλευτής στο απότερο μέλλον. Αλλά κάποιες από αυτές τις προτεραιότητες ίσως μέσα σε ένα συγκεκριμένο συντομότερο χρονικό διάστημα μπορεί κανείς να τις εξειδικεύσει. Όσο αφορά την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Access to finance Finance. Τι θα γίνει πρόθεσμα άμεσα με βήματα για να διασφαλιστεί αυτή η προσπελασιμότητα. Διαπιστώνουμε ότι οι άλλες οι οικονομίες οι και η οικονομία τη δική σα χώρα έχει, ε, έχουν προβλήματα για την ε, πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αναγκαία χρηματοδότησή του. Και βλέπουμε για την ε, αναζωογόνηση, για την βιομηχανική ανάκαμψη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι χωρί διασφάλιση τη χρηματοδότηση για αυτέ τι επιχειρήσει. Συγκεκριμένα ερωτώ, Υπάρχουν χειροπιαστά τέτοια προγράμματα και εγχειρήματα όσον αφορά το θέμα των skills, των δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τελευταία παρατήρηση, μια παράκληση θα είχα. Όχι προς το δικό μου το συμφέρον, αλλά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με ρημνό εξ ονόματος Επιτροπής, Επιτροπής για να το πω αυτό. Έχει υποβάλει ενδιαφέρουσες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτραπέζης για τη δημιουργία πλατφόρμας, πλατφορμών, δηλαδή ε, ή ας το πω έτσι ομαδοποιημένα ε, κατηγοριοποιημένων εταιριών και πρωτοβουλειών όπως για την περιφέρεια της Φλάνδρας για παράδειγμα στο Βέλγιο και βλέπω ότι υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις από το Συμβούλιο με υπονοείται η επιφύλαξη να μην αναμειγνύεται λένε οι Βρυξέλλες στα τέτοια θέματα περιφερειακά και άλλα και από πλευρά του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών κάτι τέτοιο διέγνωσα όταν γινόταν λόγο για αυτή την πολιτική παράκλησή μου βοηθήστε κύριε Υπουργέ αυτή η πολύ πραγματιστική εξειδικευμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθηθούν οι περιφέρειες να μην τροχοπεδούνται από εθνικά μικροσυμφέροντα, μικρονοϊκά συμφέροντα ότι δεν επιτρέπεται λέει κάτι τέτοιο να γίνει. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και να επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για του, την κούρα Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και Υπουργέ. σα θυμόμαστε από την εποχή που ήμασταν συνάδελφοι. Πρέπει να σας πω ότι θα έλεγα μετεπένων, σούμα κουμπλάουντε τον στόχο σας για τη, την ελληνική προεδρία και το πώς θα ορίσετε, θα ορίζετε τις προτεραιότητες της Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι ο πρώτος που θέτει την επιτροπή κατά της, που έθεσε τον, ξεκίνησε τον αγώνα κατά της γραφειοκρατίας ήταν ο αυτοκράτορας Αύγουστος. Ε, φέτος γιορτάζουμε τα 2.000 χρόνια από το θάνατό του σε όλη την Ευρώπη υποθέτω. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι στον τομέα της μάχης κατά της γραφειοκρατίας απέτυχε και αυτός και όλοι οι άλλοι μετά από αυτόν. Μέχρι και ο κύριος Στόιμπερ, ο, πρό, ο πρόσφατος πρόεδρος της Επιτροπής ε, Καταπολέμησης της Γραφειοκρατίας. Καλά, δεν συγκρίνω τον, ε, Αύγουστο, τον Τιβέριο Αύγουστο με τον Στόιμπερ, αλλά τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι ο αγώνας κατά της γραφειοκρατίας θα είναι το πιο δύσκολο καθήκον της Προεδρίας, της Ελληνικής Προεδρίας. Δεύτερο θέμα. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ο κύριος Μπιουτικόφερ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε μία έκθεση για τις μικροπιστώσεις το θυμάστε, ήσασταν ευρωβουλευτής τότε. Η μικροπίστοση είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε ένας ε, τραπεζίτης από το Μπαγκλαντές, ο Μοχάμετ Γιούνους, που επέτρεψε σε 200 εκατομμύρια άτομα ανά τον κόσμο να μετάσχουν στη χορήγηση μικρών σε μέγεθος δανείων. Εμείς εγκρίναμε την έκθεση του Κοινοβούλου, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα των ευρωομολόγων επίσης. Από την πρώτη φορά που ήρθα στο Κοινοβούλιο το 2004, είχα υπογραμμίσει την ανάγκη να υπάρχουν εργαλεία όπως τα ομοσπονδιακά ομόλογα των ΗΠΑ. Με είχαν κατακρίνει τότε διότι δεν είχαμε μια τέτοια θέση σε διεθνές επίπεδο, δεν είχαμε αυτή την αρμοδιότητα. Ωστόσο, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Έχουμε διεθνή προσωπικότητα. Άρα μπορούμε να εκδώσουμε τέτοια ευρωομόλογα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν μεγάλα προγράμματα πρωτοβουλίες στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να είσαι στην κορυφή της επιστημονικής και ερευνητικής ημερήσιας διάταξης στον κόσμο. Τρίτο σημείο, το πρόβλημα της καινοτομίας. αντιμετωπίζουμε το ζήτημα του Horizon 2020. Μια πολύ ωραία πρόταση, αλλά κατά βάση ο στόχος σε κάποια κομμάτια του προγράμματος είναι περικοπές. Προφανώς υπάρξει κάποια επέκταση σε ορισμένους τομείς, αλλά σε σημαντικούς τομείς θα αντιμετωπίσουμε μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων. Ανά την Ευρώπη πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις που έχουν καλές, πολύ καλές προτάσεις, πρωτοβουλίες, εφευρέσεις, αλλά αντιμετωπίζουν έλλειψη χρηματοδότησης. Το θέμα εκ νέου είναι θέμα πρόσβασης στην χρηματοδότηση, χρηματοδοτική κάλυψη. Η υποστήριξη ωστόσο της καινοτομία των καινοτόμων προσεγγίσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ωστόσο αμφιβολίες αν κατά τη διάρκεια των έξι μηνών θα μπορέσετε να πετύχετε κάποια πρόοδο εκεί. Διότι το γραφειοκρατικό άχθος, η ρουτίνα της γραφειοκρατίας σκοτώνει και τις καλύτερες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ τελευταία παρέμβαση από τις ομάδες, η κυρία Τζαβέλα. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στην, στα παλιά σας λιμέρια και πρέπει να πω ότι από ό,τι φαίνεται ομόφωνα όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν ότι οι προτάσεις σας για την ελληνική προεδρία είναι πράγματι πολύ σημαντικές και αποδεκτές. Ε, για να Είμαστε ρεαλιστές. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει απασχόληση και απασχόληση σημαίνει καινούργιες επενδύσεις. Αν μελετήσουμε τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία δέκα χρόνια θα δούμε ότι δεν είχαμε μία κορυφαία μεγάλη επένδυση σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει επενδυτική άπνοια στην Ευρώπη η Ευρώπη δεν είναι γοητευτική, ελκυστική για το διεθνές κεφάλαιο. Επίσης, με την κατάργηση των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων που έχουμε κάνει, γιατί επικεντρωθήκαμε όλοι σε μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Αυτή λοιπόν η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική κατήργησε στην ουσία και τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων με αποτέλεσμα να μην έχουμε παραγωγή απασχόλησης ούτε από εκεί αλλά να χάσουμε και ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης που ήταν η ποιότητα των υποδομών της. Δηλαδή μπορεί να είχε άλλα μη ελκυστικά χαρακτηριστικά η επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά τουλάχιστον οι υποδομές ήταν υψηλής ποιότητας. Τώρα το χάσαμε και αυτό. Έχουμε λοιπόν μία Ευρώπη η οποία γερνάει, η οποία δεν είναι ανταγωνιστική, η οποία μεγαλώνει μέσα σε ένα δεδαλώδες γραφειοκρατικό περιβάλλον. Έχουμε μπροστά μας δύο σύμφωνα ελευθέρου εμπορίου που προχωράν οι Ηνωμένε Πολιτείε, το ένα με την Ευρώπη και το άλλο με την Άπο Ανατολή. Η πρόβλεψή μου είναι ότι το σύμφωνο με την Άπο Ανατολή θα προχωρήσει γρηγορότερα. Και αυτό γιατί είναι πιο ελαστική από ότι είναι ο βαρύς γραφειοκρατικός οργανισμός της Ευρώπης και αυτό θα είναι άλλο ένα πρόβλημα στην ευρωπαϊκή ε, ανταγωνιστικότητα ε, άκουσα εδώ κριτική γιατί δεν προχωράμε και προέρχεται από κόμματα τα οποία όταν πάμε να προχωρήσουμε σε κάποιες τολμηρές αποφάσεις και να πάει μπροστά η Ευρώπη επικαλούμενη είτε το περιβάλλον με μια δογματική προσέγγιση είτε τα ανθρώπινα δικαιώματα πάλι με μια δογματική προσέγγιση καταργούν και εμποδίζουν κάθε προσπάθεια αναθεώρησης. Μιλήσαμε για το θέμα της υψηλής ενέργειας. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση των ενδογενών πόρων της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Έχουμε καταντήσει να εισάγουμε τα πάντα. Γιατί, Γιατί φοβόμαστε την πρόοδο, την πρόοδο στις εξορίξεις η ευρώπη δεν θα είχε φτάσει εδώ που είναι αν δεν είχε τολμηρούς άνδρες και γυναίκες οι οποίοι βλέποντας το πρόβλημα ως πρόκληση το λύσανε και προχωρήσανε. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτό είναι επώδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι επώδυνο για το περιβάλλον και να το σταματάμε θα βρούμε τη λύση βάσει των κονδυλίων της έρευνας και ανάπτυξης και θα προχωρήσουμε. αν δεν προχωρήσουμε κυρίες και κύριοι η ευρώπη πεθαίνει. ένα σημείο λοιπόν κύριε υπουργέ είναι το θέμα της αξιοποίησης των ενδογενών πόρων για την ενέργεια. το δεύτερο σημείο στην ελλάδα εσείς ο υπουργός εφαρμόσατε, κάνατε μια πολύ αξιόλογη μελέτη. βρήκατε από τον όσα ποια νομοθετήματα είναι αυτά τα οποία επικαλύπτουν το ένα το άλλο και τα οποία επιβαρύνουν το ελληνικό προϊόν και το κόστος ζωής των πολιτών. Κάτι πολύ γρήγορα που θα μπορούσατε να κάνετε με την ελληνική προεδρία είναι να κάνετε μία μελέτη για να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί νόμοι οι οποίοι επιβαρύνουν το κόστος ζωής στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τον Οκτώβριο θα έχουμε την δημοσιοποίηση των πολιτικών αρκετών τομέων για την εσωτερική αγορά. Θα μπορούσατε λοιπόν να είχατε βοηθήσει συγκεκριμένα με αυτή τη μελέτη για να μην προχωρήσουμε πάλι σε εκπόνηση πολιτικών για την ε, εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά οι οποίες θα είναι βεβαρημένες με όλο αυτό το νομοθετικό. Επανέρχομαι και λέω ότι κυρίες και κύριοι πρέπει να αναθεωρήσουμε και προσεγγίσεις και στάσεις για να μπορέσουμε να σώσουμε την Ευρώπη και τις νέες γενιές της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, τα ξέρετε όλα αυτά και θα μπορούσατε ταχύτατα και πρακτικά. Έχετε ρεαλισμό στις προτάσεις. Θα πρέπει να βρείτε και μία πρακτική προσέγγιση για να προχωρήσουν γρήγορα αυτά. Άλλωστε έχετε πικρή εμπειρία από αυτό που βλέπουμε που συμβαίνει στην Ελλάδα και το οποίο είναι αποτέλεσμα μη τολμηρών πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ας ακούσουμε τώρα τις παρεμβάσεις των συναδέλφων από τις ε, πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ συνάδελφε να τηρήσετε το δίλεπτο. Ε, δεν έχουμε χρόνο. Αν χρειαστεί να μιλήσετε λίγο παραπάνω, άντε. Ο κύριος Λάγκεν, παρακαλώ. Μάλιστα. Μπορώ ήδη να πω ότι σε σχέση με τις μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες αυτό οφείλεται στο ότι μπορούν να περιόριστα να συζητούν ε, οι συντονιστέ των μεγάλων κοινοβουλευτικών ομάδων και οι άλλοι πρέπει να περιμένουν και δεν μπορούν να παρέμβουν. Εγώ στο μέλλον, αν αγνοούνται οι κανονισμοί, δεν θα έρχομαι πλέον εδώ. Το λέω ανοιχτά. Ε, στην Οικονομική Επιτροπή περίμενα ώρε μέχρι να μπορέσω να παρέμβω και μετά παρενέβην για ένα λεπτό. Αυτέ οι μέθοδοι είναι αυτέ που οδηγούν στο να είναι ελάχιστη η παρουσία ευρωβουλευτών στην αίθουσα όπω εδώ σήμερα. Επί τη ουσία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο Χατζηδάκη έχει μεγάλη πείρα εδώ, ήταν υπουργό στην Ελλάδα, γνωρίζει πώ λειτουργούν τα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο ούτω ή άλλω και στο θεματολόγιο, στην ημερήσια διάταξη. Το τελευταίο σημείο θέλω να τονίσω ιδιαίτερα. Δηλαδή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η βιομηχανική πολιτική ω ολοκληρωμένο τμήμα τη πολιτική μα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να ε, προωθείτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Αν το πετύχετε αυτό, θα έχετε πετύχει περισσότερα από ό,τι τα 10 χρόνια τη Επιτροπή Μπαρόζο. Γιατί κατά 10 χρόνια τη Επιτροπής Μπαρόζο αυτή η ολοκληρωμένη πολιτική δεν υφίστατο και βρισκόντουσαν άλλα θέματα όπως για παράδειγμα η ε, πολιτική για το κλίμα στο προσκήνιο και όταν γινόταν η προσπάθεια για την βιομηχανική πολιτική τότε για ε, λόγους κλίματος γινόντουσαν παρεμβάσεις κλιματολογικών αλλαγών ε, και όχι για ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Αν το καταφέρετε αυτό να είναι ολοκληρωμένα άρρηκτο στοιχείο τότε θα έχετε πετύχει κάτι πολύ μεγάλο. Και το λέω αυτό και σε σχέση και με το έργο το οποίο εκτιμώ από πλευρά του κυρίου Ταγιάννη. Δεν είδα κάποια συγκεκριμένη χειροπιαστή προσέγγιση τα τελευταία πέντε χρόνια όμω από πλευρά του. Μεγάλα προγράμματα να εγκρίνονται και σχέδια. Μετά όμω ο εγω, εγωισμό των επιτρόπων για να εξευρεθούν κόκκινε διαχωριστικέ γραμμέ. Ε, Πώ προχωράμε και μετά να δαιμονοποιούνται οι Γερμανοί και να λένε ότι οδηγούν σε ανισορροπίε όσον αφορά του ε, απολογισμού. Ε, ναι, εδώ αυτέ τι προτάσει πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν δεν, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχαμε κάτι σχετικό. Είναι δύσκολη η πορεία της Ελλάδας, το ξέρουμε και συζητάμε κάθε μέρα για αυτά τα θέματα. Όμως υπάρχει μια ρύθμιση, ένας κανονισμός που τα τελευταία κατά τις τελευταίες ε, προεδρίες πάντα το ζούσα εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σε περιόδους ε, της προεδρίας τους η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση στις χώρες που είχαν, είχε αναλυφθεί η Προεδρία ήταν ενωμένε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τότε οι ε, κυβερνήσεις υποστηριζόντουσαν. Διαβάζω ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης όμως στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πρόθυμος να υποστηρίξει αυτή την κυβερνητική προσπάθεια. Θέλει μια ανατροπή, μια επανάσταση στην ε, Ευρώπη. Και τι γίνεται, υποστηρίζει η αντιπολίτευση το έργο της ε, κυβέρνησης ε, στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ. Ε, Προχωράμε με την παρέμβαση της αδερφού κυρίας Χέρτσογκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω στον κύριο Λάγκεν ότι πιστεύω ότι έχει πολλά πράγματα να κουβεντιάσει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πόσο θα μιλά και τι θα προσφέρουν, τι θα κάνουν οι επίτροποι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τέλο πάντων, αυτό θα το κάνουμε στην ε, νέα επίτροπη. Έπρεπε να το πω, δεν μπορούσα να το πω. Μία ερώτηση έχω προς τον Υπουργό. Νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα με θέματα που μπορεί να λύσει ο Υπουργό. Τα άλλα θέματα θα τα αφήσουμε για άλλη περίοδο. Μία ερώτηση έχω κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ μαζί σας ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα πρέπει να αποκατασταθεί και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος στην Ευρώπη για να δείξουμε ότι η πραγματικότητα μετράει είναι η Ελλάδα. Δεν έχουμε μόνο χρηματοοικονομική κρίση αλλά και κρίση ε, εργασία. Ό,τι βοήθεια χρειαστείτε στον τομέα αυτό είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Η ερώτηση που έχω. Έχουμε πολύ περιορισμένους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πετύχουμε αλλά υπάρχουν 23 δις στις πολιτικές συνοχής και περιφερειακής πολιτικής. Εάν κομμάτι από αυτό πάει στα προγράμματα ανταγωνιστικότητας ήταν κάτι εξαιρετικό. Έχετε κάτι υπόψη σας, σκέφτεστε πως το χτένισμα αυτών των πόρων θα μπορούσε να επιτρέψει να περάσουν στον τομέα της ανταγωνιστικότητας κομμάτι από τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει όρια στις ερωτήσεις. Η συνάδελφος, κυρία Καρβάγιο, παρακαλώ. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Υπουργέ για την περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα και για την περιγραφή των πολιτικών σας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία κατά την Προεδρία σας. Απόλυτα συμφωνώ με το πρόγραμμα το οποίο συμπεριλάβατε για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ε, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία για τους όρους που πρέπει να καλυφθούν ε, για τις επενδύσεις, ε, για την ανάπτυξη ολιστικά, σφαιρικά. Αυτή είναι η σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ωστόσο θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είμαι Πορτογαλίδα Ευρωβουλευτήνα. Στην Πορτογαλία έχουμε μια κατάσταση παράλληλη κατά κάποιο τρόπο, συγκρίσιμη με εκείνη της Ελλάδας. Ήδη κάναμε, προβήκαμε σε πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται και έχουμε μια κατάσταση κατά τους τελευταίους εννέα μήνες όπου έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές από πλευρά της Πορτογαλίας και άρχισε η ανεργία να μειώνεται. Αρχικά θεωρούσαμε ότι ήταν αυτό επίπτωση σε σχέση με την περίοδο μετά το θέρος που διακούσε μέχρι τώρα. Όμω υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε και επιδεινώνεται. Είναι η ανεργία των νέων και μάλιστα με δεξιότητες ε, και των διπλωματούχων και καταρτισμένων. Υπάρχει ε, σε σχέση με τους ιατρούς, ε, τις, ε, τους νοσοκόμους, μηχανικούς, μηχανολόγους, ε, ειδικούς για την πληροφορική που εγκαταλείπουν την Πορτογαλία και αναζητούν εργασία αλλού. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε επενδύσεις και διαμορφώνοντας ένα φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό. Η Πορτογαλία ήταν η χώρα που είχε μεγαλύτερο ποσοστό με δεξιότητες από τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Έχουμε τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό αναλογικά με τον πληθυσμό επιστημόνων και ειδικών. Μετά την ε, Δανία, τη Σουηδία, Φινλανδία ήταν η Πορτογαλία η επόμενη, τέταρτη στην Ευρώπη. Υπάρχουν επενδύσεις σε μεγάλο, ε, μεγάλη κλίμακα που γίνονται στη χώρα μας, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και οι περισσότεροι δεν πάνε στην Ευρώπη Ευρώπη. Περισσότεροι από αυτού πάνε εκτός Ευρώπης για να εργαστούν. Αυτό είναι ένα παρόμοιο πρόβλημα με εκείνο το οποίο σίγουρα εσείς αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν το οποίο κατανοείτε πάρα πολύ καλά εσείς και το γνωρίζετε. Και όχι μόνο οι χώρε αυτέ που έχουν αυτά τα προβλήματα υφίστανται το πλήγμα αυτή τη κατάσταση, κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη με κάποιε εξαιρέσει. γενικότερα λοιπόν η Ευρώπη είναι εκείνη που πλήττεται και περνά μέσα από αυτά τα δεινά. Και τι θα έπρεπε να κάνουμε θεωρείτε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αυτό το πρόβλημα και ιδιαίτερα να γίνουμε ελκυστικοί για τι βιομηχανίε μα και τι επενδύσει του. Είναι σημαντικό αυτοί οι μηχανικοί, μηχανολόγοι, άλλοι ειδικοί για, τις ε, για την πληροφορία και την πληροφορική να μπορούν να απασχολούνται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μία ερώτηση θα είχα, ένα ε, σχόλιο. Έγινε λόγος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στον ορίζοντα 2020 προσπαθήσαμε τα δημοσιονομικά από πλευράς τα κονδύλια να αυξηθούν για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποφεληθούν. Ο συνάδελφος ίσω στο Eurostar αναφερόταν αλλά γενικά έχει αυξηθεί ο προπολογισμό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτά σε σχέση με το σχόλιο του συναδέλφου. Ευχαριστούμε, κύριο Σέλμερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ καλό που ξαναβλέπουμε τον Κωστή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο συνάδελφο Λάγκη όμω είπε ότι κανεί δεν θα διαφωνήσει στην αίθουσα με αυτά που είπατε. Οπότε φοβάμαι ότι εγώ ναι θα διαφωνήσω. Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω αυτόν τον αυθαίρετο στόχο για 20% για τη βιομηχανία. Είναι μια ιδέα που κυκλοφορεί ότι, η ευρώ, ότι ένα ευρώ μάλλον από τέτοιες βιομηχανικές δραστηριότητε είναι πιο σημαντικό από ένα ευρώ που έρχεται από τον τουρισμό ή από τα δημοσιονομικά κτλ. Γιατί, να μου το εξηγήσετε αυτό. Δεύτερον, η λύση σας είναι μια βιομηχανική πολιτική. Μα το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι είχαμε πάρα πολύ βιομηχανική πολιτική. Ο κύριος Λάγκε λέει ότι χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη. Τι ωραία! Ναι, αλλά δεν θα δώσουν καμία σημασία. Τελικά χάνουμε το χρόνο μας εδώ. Προτείνω λοιπόν να λάβετε υπόψη σας τα λόγια κάποιου σοφού Αμερικανού που είπε κάποτε ότι δεν πρέπει να μάθουμε εμεί το χορτάρι να φυτρώνει, αλλά να βγάλουμε τις πέτρες από το χορτάρι. Αυτό όμως που έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα σωρό εμπόδια στη βιομηχανία, αντί να δώσουμε κίνητρα και μας κάνει εντύπωση που έχουμε πρόβλημα. Πολύ σύντομα λοιπόν θα σας πω ποια είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα το ευρώ. Μεγάλη καταστροφή που έχει κοστίσει βέβαια στην Ελλάδα πολλά, το ξέρετε εσείς, και δημιούργησε τις πιο τερατώδεις ανισορροπίες στην Ευρώπη. Και αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε, γιατί έχουμε 50% ανεργία των νέων σε κάποιες χώρε. Δεν λέω ότι έχω τη λύση. Έπειτα, υψηλά επίπεδα ρύθμιση. Αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι σε αυτά. Ναι, αλλά εσεί αντικίνητρα δίνετε στου εργοδότε και κυρίω στου μικρού. Οι εργοδότε δεν είναι πρόθυμοι να προσλάβουν. Ακούμε ότι αν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση προσλάβανε δύο παραπάνω, θα λύναμε το πρόβλημα τη ανεργία. Ε, ας τι βοηθήσουμε να το κάνουμε αντί να του βάζουμε εμπόδια στη δουλειά του. Έπειτα πολύ σωστά αναφέρεστε στο κόστο τη ενέργεια. Τεράστιο πρόβλημα και σίγουρα οδηγούνται πάρα πολλέ ευρωπαϊκές βιομηχανίες εκτός της Ευρώπης. Γιατί, Γιατί δεν έχουμε μια ενοποιημένη ενεργειακή αγορά. Χάνουμε πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων ευρώ με την αιμονή μα στι ανανόσιμε πηγέ ενέργεια και τελικά αγοράζουμε το ακριβό φυσικό αέριο από τη Ρωσία αντί να έχουμε το φθηνό άνθρακα από την Αμερική δεν θα λυθούν τα προβλήματα που αναφέρατε αν δεν αλλάξει αυτή η καταστροφική μας πολιτική. Θέλουμε μια ενωπημένη ενεργειακή πολιτική, αλλιώς δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ελπίζω αυτά τα προβλήματα να αλλάξετε, να άρετε τα εμπόδια που υπάρχουν και η βιομηχανία μόνη της θα τα βγάλει μια χαρά πέρα. Και κατά τα άλλα, συγγνώμη, πρέπει να κάνω πολύ σημαντικό τηλεφώνημα και θα προσπαθήσω, Κωστή, να είμαι πίσω για να ακούσω την απάντησή σου. Ευχαριστώ. Ε, ε, ε, δώσω τώρα το λόγο στον Υπουργό για την ανταπάντηση με μία μόνο παρατήρηση από πλευράς μου. Εκτιμήσαμε και την ρεαλιστική θέση που θέλατε να δώσετε στην παρέμβασή σας και στο πρόγραμμά σας κύριε Υπουργέ. Θα ήταν πολύ σημαντικό σε αυτή την ρεαλιστική προσέγγιση κύριε Υπουργέ να βρεθεί συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα της χρηματοδότησης και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Πρέπει να υπάρχει εξουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να μπορεί να οδηγήσει στο να φτάσουν οι χρηματοδότηση από τις τράπεζες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, διότι και εσείς έχετε τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Μανιάτη, που περιμένει ε, να, να, να σας μιλήσει. Και εγώ έχω να πάω στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, γιατί το Υπουργείο μας καλύπτει διάφορους τομείς και έχω σήμερα τρία διαφορετικά meetings στα οποία πρέπει να συμμετάσχω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιληπτικός γίνεται. Συμφωνώ με την παρατήρηση του κυρίου Λάγκε, του κυρίου Μπουτικόφα, σχεδόν όλων των συναδέλφων. Ε, συγγνώμη που λέω συνάδελφοι, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Ε, ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των λόγων και των έργων. Και ξέρετε, θα μπορούσα να πάρω το ρίσκο και να έρθω σήμερα ενώπιόν σας και να πω μέχρι τον Ιούνιο θα κάνουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θέλω να το πάρω το ρίσκο, διότι στο τέλος Ιουνίου θα γίνει ένας απολογισμός της ελληνικής προεδρίας. Και το τι θα κάνει η ελληνική προεδρία και όποια προεδρία δεν εξαρτάται μόνο από μας, μακάρι να εξαρτάται από μας. Θα εξαρτηθεί από τον κοινό παρονομαστή που θα βρεθεί μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω τόσο ανοιχτά. Αλλά είχα δοκιμάσει με συναδέλφους και με την Επιτροπή να περάσω την ιδέα ότι και εν ώψη των ευρωεκλογών ίσως θα ήταν αναγκαίο να καταλήξουμε έστω και σε ένα-δυο νομοθετικού χαρακτήρα παρεμβάσεις προκειμένου να στείλουμε το μήνυμα ότι να, νοιαζόμαστε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και δεν θα το έκανα μόνο για την ελληνική προεδρία. Προφανώς και εμείς θα είχαμε κέρδος από αυτό. Το, το, κάνουμε, θα θέλαμε να το κάνουμε συνολικά για όλη την Ευρώπη και για ένα μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και στη βιομηχανία και στους πολίτες ότι κάτι αλλάζει στην Ευρώπη. Δυστυχώς δεν φαίνεται να έγινε αυτό κατορθωτό. Έγινε κάτι άλλο κατορθωτό όμως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να είναι αφιερωμένο στη βιομηχανία, τα δύο συμβούλια ανταγωνιστικότητας να είναι και τα δύο αφιερωμένα στη βιομηχανία και να σας πω και κάτι άλλο για να μην αδικούμε όλοι τους εαυτούς μας. Ασφαλώς θα ήθελα να έχουμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο. Πολύ μεγαλύτερη πρόοδο. Αλλά επειδή θυμάμαι τι γινόταν εδώ το 2000, το 2005, το 2007, η συζήτηση τότε ήταν μόνο για το περιβάλλον. Θα μου πείτε είναι κακό να συζητάμε για το περιβάλλον. Όχι, είναι καλό να συζητάμε για το περιβάλλον, αφορά την ποιότητα της ζωής μας, αφορά το μέλλον όλων μας. Αλλά δεν είναι μόνο το περιβάλλον που έπρεπε να συζητάμε. Αγνοήσαμε τη βιομηχανία, υποτιμήσαμε τη διάσταση επιχειρηματική πολιτική και σήμερα έχουμε ανάπτυξη στην Αμερική, ανάπτυξη στην Κίνα, ύφεση στην Ευρώπη. Ε, ε, αυτό, με συγχωρείτε που θα το πω, το προκαλέσαμε και μόνοι μας σε ένα μεγάλο βαθμό άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ε, επομένως, τώρα, αν μη τι άλλο, κάπως έχουμε καταλάβει αυτό το μήνυμα και προσπαθούμε να διορθώσουμε τη ζημιά. Ελπίζω ότι οι έξι μήνες της ελληνικής προεδρίας θα συντελέσουν όσο περισσότερο γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Έρχομαι να κάνω ε, κάποιες πιο ε, συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ε, κυρία Τζόρνταν, σε σχέση με το θέμα της ενέργειας, είναι εδώ ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα και για το θέμα των CO2 emissions και για το θέμα του shale gas και όλα τα θέματα που επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της, ελληνικής της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Εγώ θα έλεγα πάλι ίσως ξεφεύγοντας από το πρωτόκολλο ότι ναι, καλώς κάναμε και πήραμε πρωτοβουλίες για το Κιώτο, καλώς κάναμε και έχουμε όλη αυτή την ευαισθησία για το περιβάλλον και στο μέλλον πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ευαισθησία για το περιβάλλον, αλλά πρέπει ε, να δούμε τι γίνεται με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, με την ανεργία, με την απασχόληση. Σας το λέει κάποιος που προέρχεται από μια χώρα που περιβάλλεται από χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια, η Τουρκία, η Βόρειος Αφρική κτλ. Ξέρετε, όποια μέτρα και αν πάρουμε εμείς σε σχέση με το περιβάλλον και τη βιομηχανία, έχουμε δίπλα μας διάφορες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θα ακολουθήσουν τους κανόνες που εμείς ακολουθούμε και επομένως βιομηχανίες μπορεί να μεταγκατασταθούν εκεί και επομένως θα έχουμε Πρώτον ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, καθώς εκείνοι θα έχουν άλλους κανόνες με βάση τους οποίους θα λειτουργούν και δεύτερον θα υφιστάμεθα τις ίδιες περιβαλλοντικές συνέπειες διότι απλώς οι βιομηχανίες αυτές θα εκπέμπουν μερικά χιλιόμετρα μακριά από εμά. Περί αυτού πρόκειται. Επομένως χρειάζεται να δούμε τα πράγματα με μια άλλη λογική και σε σχέση με τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Και με συγχωρείτε για το ότι ξεφεύγω από το πρωτόκολλο, αλλά ε, επειδή μιλήσατε έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια, με την ίδια ειλικρίνεια θέλω να σας μιλήσω ε, και, εγώ. Ε, σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τον κύριο Ράντοφ και, και, και άλλους συναδέλφους σε σχέση με, το, με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Πιστέψτε με κύριε Ράντοφ, το βιώνουμε εντονότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τα επιτόκια δανεισμού στην Ελλάδα είναι 9 και 10%. Στις ανταγωνίστριες χώρες προς την Ελλάδα είναι 4, 3, 5%. Άρα δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να είναι περισσότερο υπέρ αυτών των θέσεων από εμάς. Εμείς στην πατρίδα μας προσπαθούμε να πετύχουμε τη σταθεροποίηση, τη δημοσιονομική προσαρμογή, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας έτσι ώστε τελικώς να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της εμπιστοσύνης και αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της εμπιστοσύνης να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αλλά ε, είναι ανάγκη και η Ευρώπη να, να, αντιληφθεί και να, φαντάζομαι το καταλαβαίνει όλο ένα και περισσότερο ότι εκτός από την πολιτική αυτή της δημοσιονομικής προσαρμογής και της ε, ανταγωνιστικότητας που είναι αναγκαία υπεραναγκαία πρέπει να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα της χρηματοδότησης, επαναλαμβάνω των επιχειρήσεων, όχι με γραφειοκρατικό τρόπο. Διότι βλέπω και αντιδράσεις ορισμένων κρατών μελών, πολλών κρατών μελών, σε, ε, σε σχέση με κάποια εργαλεία που προτείνονται από διάφορους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οι αντιδράσεις είναι αρνητικές κατά το μάλλον νήτων. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε πώς σχεδιάζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ αυτά τα εργαλεία. Ε, και αυτό ε, ισχύει και για την ερώτηση της κυρίας Χέρτζοκ. Ε, δεν φτάνει να έχουμε τα όποια εργαλεία ε, στο επίπεδο του κοινοτικού προϋπολογισμού και του MFF, αλλά πρέπει να δούμε την προστιθέμενη αξία τους. Διότι καθώς έχουμε περιορισμένες χρηματοδοτικές πηγές, αυτό που έχει σημασία είναι να επενδύονται τα χρήματα με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Ε, έρχομαι σε κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό πνεύμα από την κυρία Τζαβέλα και από τον κύριο Χέλμερ. Δεν συσχετίζω το πνεύμα. Αλλά και οι δυο μίλησαν, και οι δυο μίλησαν για την ανταγωνιστικότητα και για την γραφειοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει βιομηχανική πολιτική. Δεν συμφωνούμε με τον κύριο Χέλμερ. Όχι για, να, όχι για να υποκαταστήσουμε τα κράτη-μέλη, αλλά για να υπάρχουν συνέργειες, για να υπάρχει συντονισμός, για να υπάρχει ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πιστεύουμε ταυτοχρόνως, και αυτό θα το τονίζουμε μέχρι το τέλος της Προεδρίας, ότι έχει παραγίνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με τι εθνικέ νομοθεσίε έχει παραγίνει, για να λέμε την αλήθεια, και αυτό ισχύει και για τη δική μα περίπτωση, την περίπτωση τη Ελλάδα. Αλλά χρειάζεται όντω να ξαναδούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, και ε, να δούμε πώ επιβαρύνονται οι επιχειρήσει, πώ επιβαρύνεται η βιομηχανία από αυτή την νομοθεσία. Διότι έχουμε ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα τελικώ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, όλων των αναδυόμενων αγορών με όλη αυτή την νομοθεσία υπάρχουν, υπάρχει ένα straight jacket το οποίο το έχουμε φορέσει στη βιομηχανία μας και γι' αυτό το λόγο έχουμε κυρία Τζαβέλα και την επενδυτική άπνοια στην οποία σωστά αναφερθήκατε. Και θέλω να τελειώσω με δύο παρατηρήσεις που αφορούν λιγότερο ή περισσότερο την Ελλάδα. Ε, έγιναν παρατηρήσεις από τον κύριο Λάγκεν και από την κυρία Καρβάλιο. Ε, ο κύριος Λάγκερ αναφέρθηκε στην ελληνική αντιπολίτευση, ε, η κυρία Καρβάλιο αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Σε σχέση με τη σύγκριση Ελλάδος και Πορτογαλίας, εμείς έχουμε το μειονέκτημα, κυρία Καρβάλιο, να έχουμε μια κρίση πολύ πιο οξία από ότι εσείς. Βεβαίως και εσείς έχετε τεράστιο πρόβλημα, αλλά εμείς έχουμε το πρωτάθλημα της κρίσης δυστυχώς. Έχουμε πάρει το, το πρωτάθλημα της κρίσης. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή την ώρα Έχουμε ε, το πέμπτο χαμηλότερο έλλειμμα σε όλη την Ευρωζώνη. Έχουμε πια πρωτογενές πλεόνασμα primary surplus στον, στον προϋπολογισμό μας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Ξεπεράσαμε τις προβλέψεις της Τρόικα σε σχέση με, τις, με, το τι θα κάναμε. Ο ΩΣΑ ήρθε στο Going for Growth Reports και λέει ότι είμαστε η πρώτη χώρα του ΟΣΑ σε σχέση με τις διαθωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα προβλήματα που σχετίζονται με τη ρευστότητα, access to finance, όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, και Επίσης το πρόβλημα της ρευστότητας, και ίσως αυτό ισχύει και για τη δική σας περίπτωση, συνδέεται και με το γενικότερο θέμα της εμπιστοσύνης, το confidence factor. Αυτό είναι το κλειδί, αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό εμείς ως κυβέρνηση αγνοούμε το πολιτικό κόστος και θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά όχι για να είμαστε μόνο εντάξει με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, αλλά γιατί αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον, κύριε Λάγκεν. Το πατριωτικό μας καθήκον είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ελλημάτων, του δημόσιου χρέους, της ανταγωνιστικότητας, να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα της εμπιστοσύνης, έτσι ώστε η ελληνική οικονομία, πιάνοντας το κρίσιμο σημείο, έτσι, ε, το, αυτό που λέμε we hit rock bottom, έτσι, να αρχίσει μια άλλη ε, πορεία ε, θετική προς το μέλλον. Ε, αυτό είναι που προσπαθούμε. Δεν θέλω να κάνω φυσικά κανένα σχόλιο για την ελληνική αντιπολίτευση. Ο καθένας τοποθετείται και ε, εκφράζει ε, τις απόψεις του και παίρνει και το κόστος ή το όφελος από τις απόψεις αυτές. Εμείς πάντως είμαστε αφοσιωμένοι στη δουλειά μας. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο γιατί μας το λέει η Ευρώπη, αλλά γιατί μας το λέει η συνείδησή μας. Και εκτός από αυτό σε αυτή τη φάση, στο εξάμεινο αυτό, έχουμε και την Προεδρία την ελληνική και όπως είπαμε, ο σκοπός μας είναι να έχουμε στο τέλος χειροπιαστά αποτελέσματα. Δεν έχουμε υπερφιλόδοξους στόχους, θέλουμε να έχουμε μια πραγματιστική προσέγγιση και στο τέλος, έχοντας παρουσιάσει συγκεκριμένες προτεραιότητες, συγκεκριμένους στόχους, να έχουμε πετύχει αυτούς τους στόχους. Στον κύριο Χέλμερ που ξαναγύρισε, θέλω να του πω ότι τον ευχαριστώ πολύ που ξαναγύρισε, έχασε τη μοναδική ευκαιρία να ακούσει ότι συμφωνούσα κατά 50% μαζί του. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν θα του δημιουργήσει του ίδιου ερωτήματα σε σχέση με τον προσανατολισμό του ή σε μένα, αν έχω γίνει ευρωσκεπτικιστή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ κύριε Υπουργέ για το περιεχόμενο της παρουσίασης και τις απαντήσεις σας, αλλά και για την ειλικρίνεια και τον ε, τόνο οικειότητας με τον οποίο θέλατε να συζητήσετε με την Επιτροπή μας. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα ελπίζω. <laughs> apre il ministro. Ministro Magnati. Chiede Υπουργέ Magnati. Mentre il ministro Azidakis si congeda da βγαίνει ο κύριος Χατζηδάκης, εμείς καλωσορίζουμε εδώ τον Υπουργό Μανιάτη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας που μας αφορά, που αφορά τα θέματα της δικιάς μας Επιτροπής, ιδιαίτερα το θέμα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Ακούσατε ότι ήδη τα έχουμε συζητήσει λίγο και με τον προηγούμενο Υπουργό που είχαμε εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Υπουργέ. Να ξέρετε ότι όλοι μας θέλουμε να συνεργαστούμε όσο γίνεται πιο πολύ με την ελληνική Προεδρία που βρίσκεται βέβαια σε μια κρίσιμη στιγμή. Μια περίοδο που χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Οπότε πρέπει να μετατοπίσουμε τις εργασίες μας. Σας δίνω λοιπόν το λόγο ευθύ αμέσω και επιθυμίζω στους συναδέρφους ότι Καλά έχουμε αργήσει, αλλά αργήσαμε γιατί δουλεύουμε για κανένα λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάνω έκκληση σε όλους να είναι συνθετικοί στις ερωτήσεις τους. Εσείς έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα για να μας παρουσιάσετε το έργο σας. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, ε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή να απευθύνουμε σήμερα σε εσά, σε εσά που εκπροσωπείτε το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών και ασφαλώς όλοι μαζί θέλουμε να προχωρήσουμε εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών σε μια περισσότερη Ευρώπη με περισσότερη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών και μεγαλύτερη λήψη αποφάσεων για το καλό των ίδιων των πολιτών. Ε, θα προσπαθήσω πολύ συνοπτικά να σας περιγράψω τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της ενέργειας, αλλά θεωρώ χρέος μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τις βαθιές μου ευχαριστίες για την προηγούμενη Λιθουανική Προεδρία και την προπροηγούμενη την Ιρλανδική, οι οποίες χειρίστηκαν σημαντικούς φακέλους και σε μεγάλο βαθμό προώθησαν ε, τα αντίστοιχα θέματα. Θέλω να ελπίζω ότι και η δική μας Προεδρία θα είναι εξίσου ε, επιτυχής παρά το γεγονός ότι ξεκινούμε με ένα μειονέκτημα, το μειονέκτημα ασφαλώς του λιγότερου χρόνου, των επερχόμενων εκλογών. Θέλω όμως κυρία Πρόεδρε να ελπίζω ότι ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μειονέκτημα προκειμένου να το κάνουμε πλεονέκτημα για ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Άρα ας ελπίσουμε ότι όλοι μαζί συνεργαζόμενοι στενά, Συμβούλιο, Επιτροπή και κοινοβούλιο θα βρεθούμε απέναντι στο μεγάλο δίλημα και θα απαντήσουμε με θετικό τρόπο. Επιτρέψω να σας πω ότι ουσιαστικά οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας προσδιορίζονται από τρεις ημερομηνίες ορόσημα. Τρεις προθεσμίες. Η πρώτη προθεσμία είναι μέσα στο 2014, αυτή τη χρονιά, να έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά ενέργειας. Η δεύτερη προθεσμία είναι μέσα στην επόμενη χρονιά, το 2015, να μην έχουμε κανένα κράτος μέλος που να είναι απομονωμένο από τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και εδώ περιλαμβάνουμε και τις απομονωμένες περιοχές και ασφαλώς και τις νησιωτικές περιοχές. Και η τρίτη προθεσμία ορόσημο είναι η αναμενόμενη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή του χρόνου ε, στο Παρίσι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ξεκινώ με την πρώτη προτεραιότητα που ασφαλώς είναι η προτεραιότητα να εξεταστεί η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιμένουμε σήμερα κατά σύμπτωση ε, για το πλαίσιο 2030 σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Τα πορίσματα και οι συζητήσεις που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο κείμενο θα τροφοδοτήσουν την πολιτική συζήτηση που θα κάνουμε για το ε, στο πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας του Μαρτίου και ασφαλώς θα είναι ένα πολύ καλό input για το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου επίσης. Με δύο κουβέντες, δεδομένου ότι δεν έχει νόημα να πει κανείς λεπτομέρειες λίγες ώρες πριν δημοσιοποιηθεί το κείμενο, όμως νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές πως θα πρέπει στην, ε, στο πλαίσιο ενέργεια και κλιματική αλλαγή μπροστά στο 2030 να συμφιλιώσουμε πολύ βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος ασφαλώς είναι η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Και ταυτόχρονα σε αυτό τον κεντρικό παγκόσμιο πλανητικό στόχο να προσαρμόσουμε τις εξίσου σοβαρές ανάγκες που έχουμε για την μείωση των αβεβαιοτήτων σε επενδυτές, για την μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας που κατά την άποψή μου αποτελεί ένα από τα δύο κορυφαία προβλήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνολο των προβλημάτων, ασφαλώς την ασφάλεια εφοδιασμού και βεβαίως τη βιωσιμότητα της ε, ε, ε, βιομηχανίας προκειμένου στο τέλος να έχουμε προσιτές τιμές και για τους καταναλωτές αλλά και για την ίδια τη βιομηχανία. Σημειώνω μόνο ότι η συγκεκριμένη δράση, το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι αναμφισβήτητο ότι μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα για να έχουμε μία θετική έκρηξη στα ζητήματα της καινοτομίας και της έρευνας και τεχνολογίας. Θεωρώ πως η σύζευξη των βασικών στόχων κλιματικής αλλαγής και ενέργειας μπορεί πραγματικά να φέρει μια σημαντική επανάσταση στα ζητήματα της καινοτομίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η δεύτερη προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας είναι η ανταγωνιστικότητα ε, της, ε, ε, του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι τιμές ενέργειας, χάρηκα που το συζητήσετε και με τον Υπουργό τον κύριο Χατζητάκη, αποτελεί αναμφισβήτητα μια μεγάλη πρόκληση για όλους και ασφαλώς θα είναι και ένα από τα μεγάλα θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Κορυφής του Μαρτίου. Επίσης δεύτερη, ελπίζω, θετική σύμπτωση είναι ότι σήμερα περιμένουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα για τις τιμές της ενέργειας και πώς μπορούμε να μειώσουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας όλη την ευρωπαϊκή εμπειρία, ε, τις τιμές αυτές προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Εμείς ως Ευρώπη έχουμε βιώσει την οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα έχουμε και μια μεγάλη εμπειρία στο πώς θα ξεπερνούμε επιμέρους προβλήματα. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε τον ενεργειακό μας τομέα. Άρα ξέρουμε πολύ καλά, θέλω να ελπίζω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε την αντίστοιχη εμπειρία, κοινοβούλιο, κυβερνήσεις και επιτροπή, προκειμένου να έχουμε θετικές απαντήσεις σε αυτά που συμβαίνουν στο διεθνή ορίζοντα και αναφέρομαι βεβαίως στην τελευταία επανάσταση των τελευταίων ετών στο σχιστολιθικό αέριο, στην αυξημένη παραγωγή άνθρακα από δυναμικές οικονομίες, στα εμπόδια που υπάρχουν στις αγορές φυσικού αερίου, στην υψηλή εξάρτηση που έχει η Ένωση από εισαγωγές ε, ορικτών πόρων, κυρίως φυσικού αερίου, αλλά όχι μόνο, στην ανάγκη που έχουμε για την ενίσχυση των υποδομών, στον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών που γίνεται μετά την τραγική εμπειρία του ατυχήματος στη Φουκουσίμα, στην είσοδο στο ενεργειακό μείγμα όλων των χωρών μας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έλλειψη διασυντετήρων αγωγών που πάντα αποτελεί έναν σπουδαίο παράγοντα ο οποίος προκαλεί, η έλλειψη αυτή προκαλεί πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς, στην αυξημένη φορολογία που δεν σχετίζεται με το κόστος αυτό καθεαυτό της ενέργειας, αλλά με την αυξημένη φορολογία για άλλους σκοπούς που όμως επιβάλλεται στην ενέργεια, στις ρυθμιζόμενες τιμές, στη σύνθεση των τιμών αερίου πετρελαίου, στις τιμές τις σημειακές στα χάμπ και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα απόλυτα ε, ε, προκλητικό με την θετική έννοια τοπίο μέσα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε θετικά. Να προσθέσουμε το διοικητικό βάρος που προκύπτει από πολλές και επικαλυπτόμενες και ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες και χαίρομαι που πραγματικά από την οπτική γωνία της βιομηχανίας πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, ενέργεια και βιομηχανία προκειμένου αυτό το βάρος που πάρα πολλές φορές δεν έχει καμία απολύτως λογική να μειωθεί. Να σημειώσω ότι στα ζητήματα ακριβώ της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που ως τελικό στόχο έχει στο τέλος της ημέρας να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας που έχουμε στον τομέα αυτό και να προσπαθήσουμε να τις αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας και δεν αναφέρομαι μόνον στην ενεργοβόρα βαριά βιομηχανία, αναφέρομαι εξίσου και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επίσης έχουν σοβαρό πρόβλημα υψηλού κόστου ενέργειας, το τελικό στίχημα θα πρέπει να είναι προσιτές τιμές στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι η συζήτηση που θα γίνει με την κοινωνία των πολιτών αλλά και οι δράσεις που θα αναλυφθούν από τη γόμνηνη ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη θα μας φέρει σε θετικά αποτελέσματα. Τρίτη βασική προτεραιότητα είναι ο ίδιος ο Ευρωπαίος πολίτης. Ουσιαστικά η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να χτυπήσουμε στην καρδιά του το τεράστιο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ο ασθενής κρίκος, ο κρίκος αυτός που θέλει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλους μας, που είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές. Οι ευάλωτοι καταναλωτές πρέπει να αποτελέσουν την πρώτη προτεραιότητα των στόχων μας για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Εδώ έχουμε τα εργαλεία, εκτός των άλλων, έχουμε και τα εργαλεία της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Είναι δύο στόχοι ουσιαστικά ενσωματώνονται σε μια ενιαία λογική που πιστεύουμε πραγματικά ως Προεδρία ότι θα πρέπει να πάρουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχουν μέχρι τώρα. Γιατί ακριβώς δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στα νοικοκυριά και τους πολίτες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματο. Η τέταρτη προτεραιότητα είναι ασφαλώς η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς όπως σημείωσα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας του Ιωνίου απαιτείται να έχει πολύ γόνιμη και δημιουργική τη δημόσια συμμετοχή και ασφαλώς στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε κράτη-μέλη και να χρησιμοποιήσουμε τους ενιαίους κανόνες της ενεργειακής αγοράς για όφελος των πολιτών και για ενίσχυση των περιφερειακών περιοχών, των απομονωμένων περιοχών και των νησιωτικών περιοχών. Η πέμπτη προτεραιότητα που στην πραγματικότητα αποτελεί και το βασικό θέμα συζήτησης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει στη χώρα μας 15 και 16 Μαΐου έχει τρεις επιμέρους προτεραιότητες. Πρώτον, η μελέτη, η διαφοροποίηση, η συγκεκριμενοποίηση και η ανάδειξη των εξελίξεων από την διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων μεταφοράς ενεργειακών αγαθών με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον νότιο διάδρομο και την τροφοδοσία της Ένωσης από τις πηγές της Κασπίας του Αζερβαϊτζάν σε πρώτη φάση και ευρύτερα της Κασπίας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι τελευταίες εξελίξεις, εξαιρετικά θετικές εξελίξεις στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύπρος, Ισραήλ και ελπίζουμε πολύ σύντομα και η Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν έναν νέο πόλο ε, ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης με φυσικό αέριο και πετρέλαιο και αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη και στο ευρύτερο γεωπολιτικό γίγνεσθε. Και η τρίτη προτεραιότητα του άτυπου Συμβουλίου θα είναι η συζήτηση επί της επίσπευσης και ενίσχυσης της πολύ καλής πρωτοβουλία που έχει πάρθει για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, τα περίπου 250 έργα υποδομών ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης που έρχονται να καλύψουν και με παραδοσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να προσδιορίσουμε να καλύψουν το κενό αυτό που υπάρχει σήμερα ανάμεσα σε κάθε κράτος μέλος αλλά και στη σχέση των κρατών μελών μεταξύ τους. Η τελευταία παρατήρηση και τελειώνουμε αυτό με τις προτεραιότητές μας είναι ασφαλώς η ενιοποίηση και η στήριξη των εξωτερικών σχέσεων της κοινότητας με, το, με τον εξωτερικό μας περίγυρο. Οι διεθνείς σχέσεις μας λοιπόν με ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή κοινότητα που αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο σχέσεων της Ένωσης με τις γειτονικές χώρες, οι σχέσεις μας με τη Μεσόγειο στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, η σχέση της Ένωσης με την Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και άλλες χώρες και ασφαλώς οι σχέσεις μας με τον ΑΕΡΙΝΑ, τον ΟΠΕΚ και άλλους διεθνείς οργανισμούς είναι βεβαίως ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τελειώνοντας και αφού σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, πρέπει να πω ότι με μεγάλη χαρά θα ακούσω τις ε, ερωτήσεις και θα προσπαθήσω όσο μπορώ ομαδοποιώντας να, να, να απαντήσω. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή που μου κάνετε να με ακούσετε και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για αυτή την πλούσια παρουσίαση που μας κάνετε. Θα δώσω αμέσω το λόγο στους συναδέλφους των ομάδων και μετά στους υπόλοιπους συναδέλφους. Παρακαλώ εξ αρχής να είστε σύντομοι γιατί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Η κυρία Τζόρνταν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Να ευχαριστώ τον Υπουργό κύριο Μανιάτη. Πριν είχαμε συζητήσει με τον συνάδελφό σας τον κύριο Χατζηδάκη για θέματα ανταγωνιστικότητας, αλλά επειδή η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την πολιτική ενέργεια στην αλλαγή του κλίματος ε, και περιβαλλοντικές πολιτικές είπε ότι θα απαντήσετε εσείς σε κάποιες ερωτήσει που θέσαμε. Χαίρομαι που είστε εδώ λοιπόν. Είστε υπεύθυνο και για το περιβάλλον και για την ενέργεια. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικών προτύπων. Στο παρελθόν είχα την άποψη, το αίσθημα μάλλον, ότι η ενέργεια και η ανταγωνιστικότητα ήταν κατά κάποιο τρόπο υποκείμενες πολιτικές στην αλλαγή του κλίματος και των περιβάλλον. Ποια είναι η δική σας άποψη για τη σχέση μεταξύ των διαφόρων αυτών πολιτικών. Επόμενη ερώτηση. Ενέργεια και αλλαγή του κλίματος εν ώψη του πλαισίου μέχρι το 2030. Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω ελλείψεων στην πολιτική μας για την αλλαγή του κλίματος ενώ μέχρι το 2020. Είχαμε σοβαρά προβλήματα επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, στις τιμές της ενέργειας, την επικάλυψη πολιτικών που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, την αύξηση χρήσης του άνθρακα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πού κατά την άποψή σας έγινε η τα λάθη που κάναμε και ποια λάθη πρέπει να τα βελτιώσουμε εν ώψη του πλαισίου για το 2030 και πώς. Επόμενη ερώτηση. Μιλήσατε για προμήθεια ενέργειας από την περιοχή της Κασπίας. Όπω ξέρετε, πριν από λίγες εβδομάδες... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε ότι οποιαδήποτε διακυβερνητική συμφωνία πρέπει να σέβεται τους εσωτερικούς κανόνες της, ε, τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Δύσκολο θέμα και η ερώτησή μου είναι τι, ποια πρωτοβουλία προγραμματίζεται από πλευρά Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η Τερέζα Μανδουρέλα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην Επιτροπή. Μπορείτε σίγουρα να υπολογίζετε στην μέγιστη συνεργασία μας για να προχωρήσουμε, για να προχωρήσουμε το συντομότερο εντό σε αυτό το φιλόδοξο πλήρες πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε και με, το οποίο, με τους στόχους του οποίου συμφωνούμε απόλυτα. Όπως και η προηγούμενη συνάδελφος που μίλησε και εγώ θα ήθελα να σας θέσω μία ερώτηση σε σχέση με την πρόταση του νέου πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα που θα εγκρίνει, ενέκρινε, δεν ξέρω, σήμερα το πρωί επιτροπή. Μιλήσατε σωστά για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την ασφάλεια των επενδύσεών μας. Αυτό που δεν κατάλαβα ωστόσο είναι το εξή. Ξέρετε, το ξέρετε σίγουρα ότι πριν από δύο εβδομάδες σε μια κοινή συνάντηση της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος εγκρίθηκε μια πρόταση, φιλόδοξη πρόταση που περιλάμβανε στόχους υποχρεωτικούς για τις εκπομπές αερίων διοξιδίου του, ε, ε, αερίων του θερμοκηπίου και η τήρηση των στόχων αυτών απαιτεί καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και προφανώς ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αναφερθήκατε στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα μιλώντας ε, για την εφαρμογή της οδηγίας, τα στοιχεία όμως από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, φαίνεται καθαρά ότι θα δημιουργούνταν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας αν εφαρμόζαμε σωστά αυτή την οδηγία. Το ερώτημα είναι, θα υποστηρίξει τη γραμμή αυτή το, η ελληνική προεδρία, τη γραμμή του κοινοβουλίου δηλαδή. Δεύτερον, μεθαύριο, αύριο το πρωί στην Επιτροπή, θα, θα υποψηφίσουμε μια ένσταση σε μια κατεξοδότηση πράξη για το backloading. Μπορείτε κύριε Υπουργέ να μας εξηγήσετε ή να μας ενημερώσετε για το πώς έχει κατάσταση στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Προβλέπετε να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ευχαριστώ. Για τους συντηρητικούς ο συνάδελφος Τσίσεστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις παρατηρήσεις σας. και για τις επιθυμίες που μας αναφέρατε. Τώρα, προσπαθώντας να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μερικές φορές έχουμε βεβαιότητα για το τι ακριβώς αυτό σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Σημαίνει ότι θέλουμε να αποφύγουμε, να μειώσουμε την διάσταση της κλιματικής αλλαγής ή θέλουμε να κάνουμε υπιότερες τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή, γιατί η φύση πιστεύω πάντα ότι είναι ισχυρότερη του ανθρώπου. Από την άλλη μεριά όμω, αν ακολουθήσουμε κάποια βήματα για να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε από την κλιματική αλλαγή, μου φαίνεται κάτι πάρα πολύ λογικό, μια πολύ λογική πολιτική πρόταση. Περιμένουμε βέβαια τώρα, είμαστε εν αναμονή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030. Θέλω λοιπόν εκφράσω την ελπίδα ότι το Συμβούλιο θα αποθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να έρθει με λύσεις για προβλήματα που δεν υπάρχουν ή που θα έρθει με προτάσεις στόχων που θα προβλέπουν λύσεις χωρίς να έχουμε καθορίσει προηγουμένως τους στόχους, όπως για παράδειγμα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα πολύ βασικό θέμα και αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιστεύω ότι αφήνει πίσω άλλες πτυχές της ενεργειακής πολιτικής. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ορίσουμε ποιος είναι ο στόχος μας, τι θέλουμε να πετύχουμε όσον αφορά τις εκπομπές του οξυδίου του άνθρακα ή γενικότερα αερίων του θερμοκηπίου και μετά να καθίσουμε να βρούμε τις λύσεις. Δεν μπορούμε να πούμε η λύση είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάτι ακόμα. Να ναι. Ο κύριος Χέλμετ εδώ βλέπω ότι αναθαρρύθηκε από αυτά που λέω και ζητάει και αυτό στο λόγο. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια έντονη ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Εν το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ε, ξεχνάμε την ε, ενεργειακή πολιτική. Είναι σίγουρα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά, αλλά Θέλω εδώ να εκφράσω την ευχή ότι δεν θα στρεβλώσουμε τις ενεργειακές αγορές προσπαθώντας να θεραπεύσουμε τις ενεργειακές πολιτικές. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να ε, προσέξουμε καλά. Έχουμε στρεβλώσει αρκετά τις ενεργειακές μας αγορές προς το παρόν, ευνοώντας κάποιες λύσεις όπως τις εναλλακτικές ενέργειες. Δεν πρέπει λοιπόν σε αυτές τις τρευλώσεις να προσθέσουμε και άλλες. Γιατί υπάρχει μεγάλη οικονομική απώλεια σε βάρος αυτών που ονομάζουμε ενεργειακά πιο αδύναμους, πιο ευάλωτους. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στην ε, Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Ενέργειας. Ε, μία ερώτηση έχω. Στα πλαίσια της Προεδρίας ή κατά την περίοδο της Προεδρίας ε, θα υπάρξει συζήτηση για το θέμα της εισαγωγής αερίου και πετρελαίου από τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, στα Συμβούλια Υπουργών ή στο, ε, στο συνάντηση κορυφής. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε πρώτη προτεραιότητα στα πλαίσια του Ευρωατλαντικού Συμφώνου Ελεύθερου Εμπορίου ε, ε, Ευρώπης και Αμερικής. Ε, κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους μου. Κύριε Υπουργέ, ποτέ δεν ήμασταν και ούτε είμαστε στο ίδιο πολιτικό κόμμα. Ο... Είστε ένας από τους καλύτερους υπουργούς ενέργειας που είχαμε στην Ελλάδα σε πολύ δύσκολες περιόδους. Ο τρόπος που προσεγγίζεται τα θέματα είναι και αποτελεσματικός και ρεαλιστικός και θα ήθελα να το πω αυτό μπροστά στην Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στην Προεδρία. Ε, Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων από σε ατομικό επίπεδο και είμαι βέβαιο ότι όλοι θα σεβαστείτε το δίλεπτο. Η κυρία Εντιτ Χέρτσοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Χέρτσοκ. Από την Ουγγαρία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας αναφέρατε τις προτεραιότητές σας. Σε μια πολύ δύσκολο, δύσκολη περίοδο, μια που δεν υπάρχει κάποια επίγουσα νομοθεσία που καλείστε να τελειώσετε όπως υπουργό Τηλεπικοινωνιών. Είναι δύσκολο λοιπόν για σας και επίσης επειδή σήμερα θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις μυστικές ή εν πάση περιπτώσει άγνωστες προς το παρόν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύσκολη κατάσταση για σας. Όμως, θέλω να σας πω ότι η Ελληνική Προεδρία έχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά της, γιατί μπορεί να μάθει στους Ευρωπαίους καλύτερα τι περιλαμβάνεται στις τιμές της ενέργειας. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ καιρό και εξαιτία των επιλογών που έχουμε κάνει για τις ενεργειακές πηγές, οι τιμές της ενέργειας ε, είναι τελικά ένα μυστήριο. Σε, στους Financial Times, χτες ή προχτές, διαβάσαμε με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η τιμή δεν ανταποκρίνεται στην τιμή παραγωγής. Μπορεί κανείς να δει οποιαδήποτε πηγή ενέργειας το κόστος της παραγωγής είναι χαμηλότερο στην Ευρώπη από τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ οι ενεργειακές τιμές είναι πολύ ψηλές για κάποιο άλλο λόγο. Επειδή είναι πολύ ψηλή φόρη των κρατών μελών, για παράδειγμα. Οι υπουργοί στο Συμβούλιο δηλαδή αποφασίζουν αυτές τις τιμές. Είναι Robin Hood η φορολογία αυτή στη χώρα μου, για παράδειγμα, που σκοτώνει την ανταγωνιστικότητα των ουγγρικών επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν τεχνητή δράση είναι αυτή και την κάνουν οι συνάδελφοί σας στο Συμβούλιο. Αν λοιπόν κύριε Υπουργέ μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα θα έχετε κάνει πολύ μεγάλο καλό στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και στις μελλοντικέ επενδύσεις. Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σας. Σκοπεύετε ειλικρινά να μιλήσετε με τους συναδέλφους σας για αυτό το θέμα. Ο το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Σύντομα θα θέσω δύο ερωτήματα. Κάθετος προτάσεις. Καταρχάς, υπογραμμίσατε το θέμα της αλλαγής του κλίματος και της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορεί να συνδέονται ωστόσο. Και το ΣΤΟΑ έκανε μία μελέτη που έχει να κάνει για, με την συνέργεια μεταξύ εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας που εξορισμού είναι διαδομένες σε όλη την επικράτεια και την δυνατότητα να καταστεί αποτελεσματική και η παρέμβαση χωροταξικά της ε, προσαρμογής μας στην αλλαγή του κλίματος. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεύτερο ερώτημα. ETS. Τη συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί στο Παρίσι το 2015. Πιστεύω ότι τούτο δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρξουν στοιχεία που θα χαρακτηρίζα ως κλιματικής δικαιοσύνης, δηλαδή την ανάγκη να δώσουμε πολιτική απάντηση στο πρόγραμμα του Μπαλί και την κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη των κρατών. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι η εσείς, πιστεύω ότι εσείς ανήκετε στους ηγέτες εκείνους που μπορούν να προβάλλουν τέτοιες προτάσεις στον χρόνο που, έχετε, που έχουμε στη μας μέχρι το 2015. Ευχαριστώ κυρία Βανμπρέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί έχουν υποθεί πολλά και συμφωνώ και με, τον, και με τη συντονίστριά μου, την κυρία Μαντουρέλ, που ζητάει να ακολουθήσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αποφάσεις που έχει πάρει όσον αφορά το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα 2030. Εμείς περιμένουμε σε μισή ώρα να κάνει τις προτάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως καταλαβαίνετε φοβούμαστε πολύ. Οι εφημερίδες αναφέρουν διάφορα. Η δουλειά σίγουρα είναι δύσκολη τώρα που είμαστε στο τέλος της θητείας μας και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρουμε αποτελέσματα. Να υπάρξει μια πολιτική συνένεση μεταξύ όλων και του Συμβουλίου δηλαδή για το πακέτο αυτό για το 2030. Σίγουρα υπάρχουν και θέματα ανταγωνισμού, οικονομίας κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα πακέτο τηρώντας τους στόχους οι οποίοι είναι καλοί για την οικονομία μας και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης για το σχιστολιθικό. Εδώ είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτοί που είναι υπέρ και αυτοί που είναι κατά. Πολύ έντονα όμως υπέρ ή κατά. Συμφωνούμε όμως όλοι για το ότι πρέπει, αν κάνουμε κάτι, να γίνει κάτω από τις καλύτερες δυνατόν περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε μια καλή πρωτοβουλία. Συνεπώς, μια νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να περιλαμβάνει το ότι αν υπάρξει εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου, του σχιστόλιθου, θα πρέπει αυτό να γίνει κάτω από τις καλύτερες δυνατόν προϋποθέσεις όσον αφορά το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και περιμένω την άποψή σας από αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριο Έλμερ. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη από τον Υπουργό που έχασα τις, την παρουσίασή του γιατί δυστυχώς έπρεπε να λείψω. Κάτι άκουσα όμως. Θέλω λοιπόν να πω ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και δεν υπάρχει αυτό τον αιώνα παρετέρω θέρμανση του πλανήτη. Αυτό το γεγονός και από μόνο του ε, κάνει στραβή την ε, ορθόδοξη αυτή η άποψη που λέει ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Τώρα, όσον αφορά την μείωση των ε, επιπτώσεων, αυτό σημαίνει μεγάλες δαπάνες σε μια προσπάθεια να αποφύγουμε ένα πρόβλημα το οποίο βασίζεται σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Η Μετρολογική Υπηρεσία εδώ δεν καλά καλά δεν μπορεί να μας πει αν θα βρέχει την Τρίτη όχι. Μπορεί λοιπόν να μας πει πώς θα είναι το κλίμα σε 100 χρόνια. Άρα λοιπόν βασιζόμαστε μάλλον σε ύποπτα μοντέλα, τα οποία δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε υποθέσεις. Και εξοδεύουμε δισεκατομμύρια για να καταλήξουμε μετά να διαπιστώσουμε κατά πόσο ήταν σωστές οι προβλέψεις αυτές ή όχι. Ανεξάρτητα λοιπόν τις απόψεις που έχει κανείς για την κλιματική αλλαγή, τα πακέτα που εγκρίνουμε σήμερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποδίδουν. Αυξάνουν το κόστος μόνο, διότι τελικά μάλλον αναποτελεσματικότητα προσθέτουμε. Η ενέργεια δηλαδή που πιστεύει κανείς ότι με τις εναλλακτικέ μορφές ενέργειας και η απόδοση που νομίζουμε ότι θα έχει αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. Σήμερα στον κόσμο αναπτύσσονται νέα εργοστάσια Όσου λοιπόν συσσωρευτές ηλιακή ενέργειας, ό,τι άλλη ηλεκτρική ενέργεια και τα λοιπά θα κάνουμε, η τάση του να έχουμε διοξίδιο του άνθρακα δεν πρόκειται να σταματήσει, γιατί νέα εργοστάσια που χρησιμοποιούν τον άνθρακα χτίζονται συνέχεια. Να σας υπενθυμίσω επίσης τα πρόσφατα σχόλια του Αντώνιο Ταγιάννη, η Επίτροπος υπεύθυνο για τη Βιομηχανία, που είπε ότι στην Ευρώπη φτιάχνουμε μία βιομηχανική σφαγή με τις ενεργειακές τιμές. Τι θα κάνετε εσείς για να την αποφύγουμε αυτή την βιομηχανική σφαγή. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις, πολλές παρατηρήσεις κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους, εγώ ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τους συναδέλφους ευρωβουλευτές για τις ε, ερωτήσεις και να πω ότι ε, είναι πολύ δημιουργικό για μια προεδρία όταν ξεκινά να ακούει από τους ε, ευρωβουλευτές τους προβληματισμούς, τις αγωνίες και ουσιαστικά τις προτάσεις για βελτίωση των πολιτικών της Ένωσης σε θέματα τόσο σημαντικά όσο είναι η ενέργεια, αλλά αναμφισβήτητα συνδεδεμένη με την ενέργεια και η κλιματική αλλαγή. Εγώ τώρα με την ιδιότητα ταυτόχρονα και του Υπουργού Περιβάλλοντος και του Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Ενέργειας έχω το καθήκον μαζί με και άλλους υπουργούς σε άλλα κρατημέλη να βρούμε συμβατότητες ανάμεσα σε επιλογές που καταρχήν και νομίζω όχι πολύ σωστά αρκετές φορές δείχνουν αντικρουόμενες. Διότι εδώ πρέπει να σας ξεκαθαρίσω την άποψη όχι πια της Προεδρίας η οποία οφείλει να είναι ουδέτερη και να έχει ως στόχο την εξέβρεση συμβιβαστικών λύσεων, αλλά να πω μία προσωπική άποψη. Εγώ θεωρώ ότι μπορούν ταυτόχρονα στον πλανήτη Γη να υπάρχουν και οι πολιτικές για την μείωση της κλιματικής αλλαγής και οι πολιτικές για την μείωση του ενεργειακού κόστους στα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι που είναι αναμφισβήτητο. Στόχος όλων των κοινωνιών, όλων των συμφωνιών των Ηνωμένων Εθνών είναι η θερμοκρασία του πλανήτη να μην αυξηθεί πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, πηγαίνουμε δυστυχώς, τα νέα δεν είναι ευχάριστα, με 3,6 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν το διπλάσιο από ό,τι θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο οι αναπτυγμένες οικονομίες, για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και οι ραγδαία αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, άλλες οικονομίες, και το σύνολο ουσιαστικά του πλανήτη να έχει υπόψη ότι αυτό είναι μπροστά μας. Και άρα θα πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στη συγκεκριμένη πρόκληση. Συνοψίζω λοιπόν και λέω ότι είμαι απολύτως βέβαιος πως υπάρχουν κοινέ δράσεις συμβατότητες στην επίτευξη και των δύο στόχων. Δηλαδή, μείωση των αρνητικών εξελίξεων της κλιματικής αλλαγής σε κάτω από δύο βαθμούς Κελσίου τα επόμενα πολλά χρόνια, ταυτόχρονα παραγωγή νέου πλούτου, ο οποίος να μοιράζεται δίκαια στις κοινωνίες και κυρίως στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά και τους πολίτες. Βεβαίως βασική παράμετρο σε αυτό είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να γίνει και σε πράσινες δραστηριότητες, σε δραστηριότητες αηφορίας και βιωσιμότητας, αλλά και σε παραδοσιακές δραστηριότητες. Έρχομαι λοιπόν προσπαθώντας να απαντήσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά. Ε, ε η κυρία Τζόρταν, αλλά και αρκετοί, ε, και η κυρία Τερέζα Μανουέλα και άλλοι σας, βάλατε το ζήτημα του πώς θα πρέπει να βαδίσουμε εν ώψη της αναμενόμενης σε λίγες ώρες ανακοίνωσης Επιτροπής για το κλίμα 2030. Δεν θέλω ως Προεδρία να τοποθετηθώ σε ένα κείμενο που ακόμη δεν έχει δει κανένας μας. Όμως πιστεύω πως το κείμενο αυτό με την δημιουργική συζήτηση που θα γίνει και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μπορεί πραγματικά να καταλήξει σε κάτι που θα συνιστά ελπίδα, προοπτική και όραμα και για τις κοινωνίες και για τους επενδυτές και για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη χωριστά. Πληροφορίες έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Θέλω να αποφύγω να σχολιάσω πληροφορίες. Ως προεδρεύων είναι βέβαιο ότι θα απαντήσω και θα, χαρώ να τα πούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα με την Επιτροπή σας. Όμως νομίζω ότι ε, είναι αναμφισβήτητο πως η Ένωση πρέπει να απαντήσει στην διπλή πρόκληση. Ταυτόχρονα να συνεχίσει να είναι η πρωτοπόρος διεθνική οντότητα σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και μαζί με αυτό να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που είναι σε πολύ κακό στάδιο. Απαντώ στο ζήτημα για την Κασπία και τις ε, σχέσεις που πρέπει να διέπουν ε, την Ένωση. Η Κασπία αποτελεί μια νέα ελπιδοφόρα πηγή τροφοδοσίας της Ένωσης με φυσικό αέριο κυρίως. Οι συνομιλίες που έχουμε κάνει με τον Επίτροπο, τον κύριο Έτιγκερ, διότι και ως Ελλάδα έχουμε βιώσει τα πρώτα στάδια αυτής της νέας εταιρική σχέσης που πρέπει να υπάρχει, είναι ότι από τη στιγμή που ένα κράτος μέλος κινείται στο πλαίσιο των προδιαγραφών του τρίτου ενεργειακού πακέτου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν καθυστερήσεις. Άρα αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να υπάρξει μια εξέταση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, όμως είναι αναμφισβήτητο ότι όταν έχουν ακολουθηθεί όλες οι ανάλογες, οι πρέπουσες διαδικασίες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερούν. Και ο, ο Επίτροπος συμφωνεί σε αυτό και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας. Θέλω να κάνω ένα ιδιαίτερο σχόλιο για τα ζητήματα. Επιτρέψτε μου να πω, θεωρώ ότι ο πιο παραμελημένος και αγνοημένος παράγοντας και στο επίπεδο των, της δημόσιας και στο επίπεδο των επενδύσεων και στο επίπεδο των εθνικών πολιτικών στα ζητήματα ε, της ενέργειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Σας το λέω και με την ιδιότητα του Υπουργού που είναι αρμόδιος για το αστικό περιβάλλον και τον τρόπο καθημερινής διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών η πρόκληση μπροστά μας, κυρίως για τις χώρες του Νότου, αλλά όχι μόνο για τις χώρες του Νότου, είναι η μέσα από την ενεργειακή θωράκιση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Σε όλη την Ευρώπη έχουμε χτίσει πολλά σπίτια. πρώτα κατοικίες και δεύτερες κατοικίες. Σε πάρα πολλές χώρες όμως με πολύ μικρή ενεργειακή θωράκιση έχοντας μπροστά μας την πρόκληση της ανεργίας στον τομέα της οικοδομής, της υποβάθμισης του επίπεδου καθημερινής διαβίωσης των νοικοκυριών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος και της ανάγκης να δώσουμε όθηση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης που έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, η προσωπική μου άποψη, αν μπορώ να την καταθέσω, είναι ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα τόσο στον τομέα της κατοικίας, όσο και στον τομέα των δημοσίων και των επαγγελματικών κτηρίων, αλλά και των μηχανημάτων, αποτελεί μια τεράστια αναπτυξιακή πρόκληση, στην οποία η Ένωση, όλοι εμείς, πρέπει να απαντήσουμε πολύ επιθετικά, πολύ θετικά, με δημιουργία θέσεων εργασίας, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων και με μία προοπτική να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο. σχιστολιθικό αέριο. Έχει τεθεί και από την κυρία Τζαβέλα και την... σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι λίγο ε, υπερβολικά, αλλά ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Ε... Και από την κυρία Βαν Μπρέμπ και από άλλους συναδέλφους. Η Επιτροπή αποφάσισε για το σχιστολιθικό αέριο να βγάλει recommendations μόνο συστάσεις. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στα συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος ο προβληματισμός είναι έντονος. Είναι λιγότερο έντονος ο προβληματισμός στα συμβούλια των Υπουργών Ενέργειας. Άρα έχουμε πολλαπλούς διαλόγους όχι μόνο στο επίπεδο των θεσμών της κοινότητας αλλά και μέσα στο, στο, στο εθνικό επίπεδο κάθε κράτος μέλος. Και ασφαλώς έχουμε στην ίδια την κοινωνία των πολιτών. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας κάτι. Ότι το σχιστολιθικό αέριο είναι μια σύγχρονη, μια καινούρια μάλλον τεχνολογία, η οποία έχει αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερη παρατήρηση ότι η Ευρώπη έχει τα δικά της ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο κατοίκησης που είναι εξαιρετικά πιο πυκνός, είναι πιο πυκνοκατοικημένη η Ένωση της Ηνωμένες Πολιτείας και ασφαλώς ότι αυτό που μπορεί να συνιστά μια διέξοδο για φθηνότερη πρώτη ενεργειακή ύλη δεν μπορεί παρά πάντα να παντρεύεται με τους αυστηρότατους περιβαλλοντικούς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουμε. Το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει διαμορφωσεί άποψη. Θα περιμένουμε πραγματικά τις, τον τρόπο προσέγγισης που θα γίνει από την ε, ανακοίνωση της Επιτροπής. Ε, είμαι προετοιμασμένος για πολύ θερμές συζητήσεις, πολύ έντονες συζητήσεις στο πλαίσιο και των δύο Συμβουλίων, και του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Πιστεύω όμως ότι η οι ηγέτες των κρατών μελών μας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κορυφής μέσα στο Μάρτιο θα δώσουν και αυτή τις αντίστοιχες ε, κατευθύνσεις. Η κυρία Χέρτσοκ έκανε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Έχω ε, λίγο δεν έχω. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Για το τι σημαίνει ενεργειακό κόστος. Και θεωρώ ότι σε πάρα πολλές χώρες γίνεται μια σύγχυση. Συγχαίουμε το κόστος της ενέργειας με τα χρήματα που πληρώνει ο πολίτης όταν του έρχεται ο λογαριασμός της ενέργειας. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο πολίτης έχει πλήρη απεικόνηση του πόσο είναι το καθαρό ενεργειακό κόστος και πόσα είναι οι φόροι που επιβάλλουν τα Υπουργεία Οικονομικών, τα τέλη που έρχονται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, άλλοι φόροι και τέλη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους να είναι απόλυτα σαφές στο λογαριασμό που πληρώνει ο πολίτης, είτε ο πολίτης είτε η βιομηχανία, να είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το πραγματικό κόστος της ενέργειας και ως προς την παραγωγή, το ανταγωνιστικό κόστος και ως προς την μεταφορά το ρυθμιζόμενο κάθε φορά κόστος και ποιο είναι το εξωτερικό της ενέργειας κόστος. Άρα, συμφωνώ με την παρατήρηση, έχουμε βαθιά ανάγκη να ξεκαθαρίζουμε σε όλες τις χώρες ε, ποιο είναι το κόστος. Και να τελειώσω με τον κύριο Χέλμερ, ο οποίος έκανε και την τελευταία ερώτηση, να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τις απόψεις των ανθρώπων που ε, πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ανθρωπογενής παρέμβαση στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγή. Οφείλω να σα πω όμως ότι διαφωνώ απολύτω θεωρώ ότι η ανθρωπότητα με τον τρόπο που λειτουργήσε έχει επιφέρει τεράστιες βλάβες. Ε, μου έδωσαν ένα στατιστικό στοιχείο τις προηγούμενες μέρες ε, δημοσιεύτηκαν μέσα το 2013 το λέω με κάθε σεβασμό σε όλες τις απόψεις γιατί έτσι πρέπει να γίνεται δημοσιεύτηκαν μέσα το 2013 περίπου 3.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και το 99% των επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα ασπάζονται την άποψη ότι η ανθρωπότητα, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας εκτός από τις φυσικές ε, συνθήκες. Η ίδια η, οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος επιβαρύνει το περιβάλλον και άρα εδώ έρχεται η υποχρέωση των κοινωνιών να αναστρέψουν αυτή την πορεία. Προσπάθησα να απαντήσω κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σα. ελπίζω να μην μακρηγόρησα και ελπίζω να απάντησα όσο καλύτερα μπόρεσα στις ερωτήσει των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαστε όλοι εξαιρετικά ικανοποιημένοι από αυτή την πρωινή σειρά συναντήσεων και από τη δική σας παρέμβαση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. accogliamo il ministro Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και να του ζητήσω συγγνώμη καταρχάς για την καθυστέρηση που οφείλεται στο ότι οι παρεμβάσει των συναδέλφων, οι συζητήσει με του συναδέλφου σα ήταν τόσο ενδιαφέρουσε που. Μισό, μισό. Δεν υπάρχει διερμηνία. Έλεγα, ζητούμε συγγνώμη από τον Υπουργό για την καθυστέρηση και του δίνω μέσω το λόγο ευχαριστώντας τον για την παρουσία του εδώ είναι υπουργό με πολλέ αρμοδιότητε. Αυτό που μα ενδιαφέρει στη δική μα αρμοδιότητα είναι η έρευνα. Άρα του ζητώ να πάρει το λόγο για τον χρόνο που θεωρεί αναγκαίο και κατόπιν θα ακούσουμε τι παρεμβάσει των συναδέλφων και την ανταπάντηση. Και πάλι συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλίμονο, κανένα πρόβλημα κυρία Πρόεδρε, ίσα ίσα όταν υπάρχει μια πολύ καλή συζήτηση. No? No? We'll wait for a couple of seconds, okay. Να παρακαλέσουμε τους υπεύθυνους των υπηρεσιών διαμηνίας να τσεκάρουν ότι λειτουργούν όλες οι καμπίνες. Η ελληνική καμπίνα ακούγεται ωστόσο, έτσι. Ακούτε την ελληνική καμπίνα. Ναι. Ωραία. Not yet. Should I switch to English? <laughs> ça marche, ça marche maintenant. Il dit que ça marche Οκ. prego. Ok. Ok. Οκ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κυρία Πρόεδρε, ίσα ίσα όταν υπάρχουν ε, ενδιαφέρουσες συζητήσεις είναι πολύ θετικό και θα ήθελα καταρχήν ε, κυρία Πρόεδρε Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, να πω εξ αρχής ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μπροστά. Πρόβλημα διερμηνίας. Να παρουσιάσουμε τις ε, προτεραιότητες ελληνικής προεδρίας για τις πολιτικές... Ε, la prego, <laughs> sorry. There is something that doesn't work. Cosa voglio fare questo? Τώρα ακούγεστε. Όχι, μπορείτε... δεν Possiamo cercare di capire che e Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το σύστημα. Έλεγα ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας για να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για τις πολιτικές έρευνας πολιτικές καινοτομίας αλλά και του διαστήματος. Και στο εξάμεινο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούμαστε σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας να υλοποιήσουμε τους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Και καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ιρλανδική και την ε, Λιθουανική Προεδρία, όλα τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεργασία που είχαμε στην προετοιμασία, αλλά βεβαίως και για το σημαντικό, το αξιοθάμαστο θα έλεγα έργο που παρήχθη κατά τη διάρκεια του 2013 και το οποίο μας επιτρέπει να εργαστούμε ως ελληνική προεδρία στην υπηρεσία των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, με την ε, ανεργία να φτάνει σε ιστορικά υψηλά, σε πολλά κράτη-μέλη, και μια ανεργία η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους και βέβαια την ύφεση να απειλεί πάντοτε τις ε, ευρωπαϊκές οικονομίες, η ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για όλους, πρωταρχικής σημασίας για την Ευρώπη, πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Προεδρία, στο σύνολο βέβαια των θεματικών δράσεων της. Και η ανάπτυξη είναι η μόνη απάντηση στην κρίση, γιατί η ανάπτυξη δημιουργεί θέσει εργασίας, η ανάπτυξη εδραιώνει την πολιτική σταθερότητα, ιδιαίτερα σε χώρες που κλειδονίζονται από την κρίση. Η ανάπτυξη διορθώνει κοινωνικές ανισορροπίες και ανισότητες. Η ανάπτυξη ενισχύει την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Και όλοι γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται εμένα να το πω σε αυτή την αίθουσα, ότι η συμβολή της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη είναι καταλητική. Και αυτό τεκμηριώνεται και από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020, σύμφωνα με τους οποίους γνωρίζουμε ότι η επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία, εάν φτάσει το ποσοστό του 3% σε έναν ευρωπαϊκό μέσο όρο μέχρι το 2010, μπορεί να μας αποφέρει μέχρι και 3,5-3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ως το 2019. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η διεθνής τώρα διάσταση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας παραμένει ένα σημαντικό στοιχείο, ένα σημαντικό σημείο στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας που σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο 2014 για να πραγματοποιηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτομία. Και ειδικότερα θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση της κινητικότητας, για τη βελτίωση της κινητικότητας των προοπτικών της σταδιοδρομίας των ερευνητών μας, για τη βελτίωση της κινητικότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών μας, για την ελκυστικότητα της Ευρώπης για τους ξένους ερευνητές. Και θεωρούμε ότι μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και όλων των εμπλεκομένων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο αλλά και προϋπόθεση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Υπό το φως των σημερινών δύσκολων δημοσιονομικών ζητημάτων όλες οι δαπάνε για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και την καινοτομία πρέπει να είναι στοχοθετημένες, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ώστε έτσι να πετύχουμε μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, των ευρωπαϊκών οικονομιών. Και οι επενδύσεις αυτές στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν να μετατραπούν σε εμπορεύσιμα προϊόντα, σε υπηρεσίες, και έτσι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ανάπτυξης, στη δημιουργία απασχολήση, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η Ένωση καινοτομία είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μετατρέψει την Ευρώπη σε ένα φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον. Και γι' αυτό χαιρετίζουμε την προσπάθεια που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον ΩΣΑ για την ανάπτυξη ενός δίκτυ καινοτομία για την Ευρώπη του 2020 που αναμένεται να έχει σοβαρές και σημαντικές συνέπειες. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιηθεί η πολιτική ορίζοντας 2020, Horizon 2020, από τις αρχές του 2014 και να αναδείξουμε τον καταλητικό ρόλο της πολιτικής αυτής για την ανάπτυξη και τη συμβολή της πολιτικής αυτής στη δημιουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας του μέλλοντος αλλά και τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς καλούμεθα να ολοκληρώσουμε το πακέτο καινοτομίας, το οποίο, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, περιλαμβάνει εννέα νομοθετικές πράξεις, με τις οποίες θα συσταθούν ή θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τέσσερις μεγάλες συμπράξεις δημοσίου-δημοσίου και πέντε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Με αυτές τις συμπράξεις αναμένεται η Ευρώπη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε τομείς αιχμής και να δημιουργηθούν και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τομείς όπως βιομηχανίες βιολογικής βάσης, τα καινοτόμα φάρμακα, οι κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου, η αεροναυτική τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα, μετρολογία, ενεργός και υποστηριζόμενη διαβίωση, οι κλινικές δοκιμές, το πρόγραμμα για τις ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, στοχεύουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτηση σύμπραξης δημόσιο ιδιωτικού τομέα για τις αερομεταφορές, το ΣΕΖΑ. Και αναμένουμε βέβαια στην ψήφιση του πακέτου από την Επιτροπή αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους παράγοντες και όλους τους εμπλεκόμενους του Κοινοβουλίου με τους οποίους έχουμε ήδη ξεκινήσει άτυπες συναντήσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή αυτών των συζητήσεων, αυτών των διαπραγματεύσεων. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Προεδρία, η Ελληνική Προεδρία, ανταποκρινόμενη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα οποία ζητήθηκε η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η ενδυνάμωση της διαδικασίας ελέγχου, της προόδου αν θέλετε για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, προτίθεται να υποβάλει στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Φεβρουαρίου μια πρόταση για την υιοθέτηση των σχετικών συμπερασμάτων. Πέραν όλων των φακέλων που προαναφέραμε και για τους οποίους θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι απόλυτη, συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα για μας, η ελληνική προεδρία σε συνεργασία και με τη στήριξη κρατών μελών και κυρίως θα έλεγα από την περιοχή της, Νοτι... της Νότιας Ευρώπης θέλει να ξεκινήσει έναν διάλογο, έναν πολιτικό διάλογο για μια ευρωμεσογειακή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας προσδοκώντας να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ενδεχομένως στη βάση του άρθρου 185 της συνθήκης. Είναι ένα όραμα, αν θέλετε, που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια και θεωρούμε ότι σιγά σιγά οριμάζουν οι συνθήκες για να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του. Και αυτό το θέμα θα αποτελέσει και ένα βασικό σημείο της πολιτικής συζήτησης κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου το Μάιο του 2014. Επίσης, θα συνδράμουμε στην εμβάθυνση των ζητημάτων καινοτομία του δημοσίου. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αναλυθούν επιπλέον πρωτοβουλίες για την ανάδειξη αλλά και την εξειδίκευση αυτού του σημαντικού ζητήματος. Όσον αφορά την ε, πολιτική του διαστήματος, τα διαστημικά συστήματα μας δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογών ευρέως φάσματος που γνωρίζουμε όλοι ότι διαδραματίζουν έναν σημαντικό, ένα θεμελιώδη ρόλο στην καθημερινότητά μας. Τηλεόραση, το διαδίκτυο, η πλοήγηση, η μετεωρολογία. Η πολιτική λοιπόν του διαστήματος είναι ένα εργαλείο, ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτών μας, στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, μας, οι πολιτικές που συνδέονται είναι πολιτικές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, με την κρατική και ιδιωτική ασφάλεια, με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, με τις μεταφορές, με την κοινωνία της πληροφορίας. Αποτελεί το διάστημα, θα λέγαμε, γεννήτωρα γνώσεων, γεννήτωρα νέων προϊόντων, νέων μορφών βιομηχανικής συνεργασίας αποτελεί κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και θα λέγαμε ότι είναι και στρατηγική σημασίας για την, για την παγκόσμια σκηνή. Γι' αυτό λοιπόν το, έχουμε το πρώτο μισό του 2014 που βλέπουμε από ευρωπαϊκής πλευράς το δυναμικό ξεκίνημα σημαντικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το, το διάστημα, τον Καλλιλέο, τον Κοπέρνικους, συμπεριλαμβανομένων των ε, αναμενόμενων εκτοξεύσεων του πρώτου δορυφόρου τηλεσκόπησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και περαιτέρω δορυφόρων του συστήματος Γκαλιλαίου. Και η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων είναι σημαντική για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο για την κατασκευή διαστημικών υποδομών, όσο και για την χορηγία υπηρεσιών, αλλά και για την ανάπτυξη εφαρμογών. Και στηρίζεται βέβαια όλη η πολιτική αυτή σε μια στενότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Επίσης ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και έχει καταστεί μείζονος σημασίας είναι η προστασία των διαστημικών υποδομών για τον μετριασμό κινδύνων σύγκρουσης είναι απαραίτητο να εντοπίζονται, να παρακολουθούνται δορυφόροι και διαστημικά υπολείμματα, να καταχωρούνται οι θέσεις τους, να παρακολουθούνται οι κινήσεις τους και όταν βέβαια ενέχεται μια πιθανότητα, ένα κίνδυνο σύγκρουσης, να προειδοποιούνται οι φορείς διαχείρισης δορυφόρων, να μετακινούν τους δορυφόρους και ούτε καθεξής. Αυτούς τους στόχους καλείται να καλύψει η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την επιτήρηση και την παρακολούθηση του διαστήματος, οι τροποποιήσεις της οποίας άλλωστε έχουν ε, ψηφιστεί από την Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου. Οι δικές μας προτεραιότητες, οι προτεραιότητες της Προεδρίας για την πολιτική διαστήματος έρχονται να, να ενισχύσουν όλα αυτά, μια και επικεντρώνονται στους κάτω τρει άξονες. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης του προγράμματος Κοπέρνικους, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του πλαισίου στήριξης, επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος, το Space Surveillance and Tracking, και την περαιτέρω ανάλυση του πλαισίου συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σχετικά με τον πολιτικό στόχο για την ολοκλήρωση του νομοθετικού φακέλου του πλαισίου Space Surveillance and Tracking, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι τα κράτη-μέλη ήδη εξουσιοδότησαν την Προεδρία να ξεκινήσει τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις και ότι η διαδικασία των άτυπων τριλόγων έχει ήδη ξεκινήσει. Και εργαζόμαστε με εντατικό ρυθμό ώστε να ολοκληρώσουμε αυτά τα ζητήματα μέσα στα απαραίτητα χρονικά πλαίσια και θα ήθελα για άλλη μια φορά εδώ να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους γιατί υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όπως ήδη ανέφερα, αποτελεί για μας πολιτική προτεραιότητα ο μη νομοθετικός φάκελος, ο φάκελος που δεν έχει νομοθετική ε, πρωτοβουλία, των σχέσεων της Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, όπως προβλέπονται από τη συνθήκη. Και η σχέση αυτή καθορίζεται από το άρθρο 189 της συνθήκης, ενώ γνωρίζουμε ότι το υπάρχον σύμφωνο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών θα λήξει το 2016. Και εξειδικεύοντας αυτήν την προτεραιότητα, η Προεδρία προτίθεται να οργανώσει μια ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Φεβρουαρίου, καθώς και μια άτυπη πολιτική συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματος του Ιδίου Συμβουλίου παρουσία του Γενικού Διευθυντού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, του κ. Ντοντέν. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συμπεράσματα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Μαΐου. Για το φάκελο αυτό θα συνεργαστούμε, συνεργαζόμαστε ήδη στενά με την επόμενη Προεδρία, την Ιταλική Προεδρία, προκειμένου να έχουμε ένα κοινό σχέδιο δράσης του Συμβουλίου για το 2014 και το οποίο να μπορέσει να τροφοδοτήσει τις μελλοντικές προτάσεις Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή της συνθήκης. Τέλος, θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι πέραν των πολιτικών πρωτοβουλειών σε επίπεδο Συμβουλίου, η Ελληνική Προεδρία έχει προγραμματίσει περίπου 12 εκδηλώσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και ενδεικτικά θα αναφέρω ότι για την πολιτική έρευνας και καινοτομίας έχουμε το Διεθνές Συνέδριο για τις Ερευνητικές Υποδομές, το Συνέδριο για την Διεθνή Ερευνητική Συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις χώρες του έξινου πόντου και για την πολιτική του διαστήματος έχουμε το Συνέδριο Κοπέρνικου στο οποίο συμπίπτει με την εκκίνηση του προγράμματος για την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου Sentinel αλλά και το Συνέδριο για την Ασφάλεια και το Διάστημα. Και επίσης, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, κάναμε μια ε, εκδήλωση στην Αθήνα για την έναρξη του Horizon 2020 που έγινε την επόμενη μέρα από τη Σύνοδο του Κολεγίου των Επιτρόπων στις 10 Ιανουαρίου που μας πέρασε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό και την Επιτροπή για την ε, βοήθεια και τη συνεργασία για, όλων, για, την διοργαν... για όλες αυτές τις διοργανώσεις αλλά και να, ε, ε, να ενημερώσω ότι θα υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση και οι προσκλήσεις προς τα μέλη του Κοινοβουλίου και την Πρόεδρο των Επιτροπών, της Επιτροπής όσον αφορά αυτήν, αυτές τις εκδηλώσεις και φυσικά θα είναι για μας ιδιαίτερη τιμή να παραστείτε σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η Ελληνική Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να έχουμε μια επιτυχή ε, διεκπαιρέωση όλων των ζητημάτων κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτω ώστε να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο τους κοινούς μας στόχους. Και ευελπιστούμε για μια συνεχή και επικοδομητική συνεργασία με τα κράτη-μέλη, την Επιτροπή αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε τη μεριά μας για την δυναμική εκκίνηση του μεγαλύτερου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Horizon 2020, αλλά και του Κοπέρνικους και του SST και να βάλουμε το θεμέλιο για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων για τα χρόνια που έρχονται. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την πλούσια παρουσίασή σας. Θα ζητούσα από τους συναδέλφους να είναι πραγματικά συνθετικοί στα δύο λεπτά για να μπορέσει ο υπουργό να απαντήσει στις παρεμβάσεις σας. Η κυρία Καρβάλιο ξεκινά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και εξ ονόματος του ΕΡΚ σας καλωσορίζουμε εδώ ανάμεσά μας σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα οποία μας δηλώσατε ως κύριες προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας ευθυγραμμίζονται απόλυτα και με τις δικές μας προτεραιότητες και αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει στις, ε, και κατά τη γνώμη μας η δική σας παρουσία στην Προεδρία σας θα είναι κέρια σημασία. Σε, σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία ξεκινά η υλοποίηση πολύ σημαντικών προγραμμάτων και σχεδίων και είναι ωραίο αυτό και είναι πολύ θετικό. Καθένας κάνει λόγο για αυτά όταν τα εγκρίνουμε αυτά τα προγράμματα, αλλά οι λεπτομέρειες υλοποίησης της πρώτης εφαρμογής και υλοποίησης είναι πολύ σημαντικές υποθέσεις και υπάρχει μεγάλη ευθύνη από πλευράς του Συμβουλίου, διότι θα είναι μια μεταβατική περίοδος και για το Κοινοβούλιο αυτή, για μας. Έχετε πολύ σημαντικό έργο λοιπόν ενώπιόν σας, για παράδειγμα για να δώσετε συνέχεια, follow-up και να μεριμνήσετε πώς θα εφαρμοστεί ο χρονορίζοντας 2020 ως εγχείρημα. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό το στόχο και το αποτέλεσμα του ως στόχου, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν και πράγματα όπως η απλούστευση για παράδειγμα, πρέπει να υλοποιηθούν, όλα να γίνουν πιο διαφανή. Όλα αυτά είναι αρχές που εγκρίναμε και υπερψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διεύρυνση του πλαισίου συμμετοχής, η εμπλοκή και συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πόσο χρονορίζοντας 2020 θα μπορέσει να βοηθήσει και να αυξήσει την απασχόληση των νέων, νέων ανθρώπων με δεξιότητες και ικανότητες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα παρακολουθήσετε και να εφαρμοστούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσετε γι' αυτό. Δεύτερη προτεραιότητα, η κατηγορία της Ευρωπαϊκής Έρευνας και της ε, επιστήμης και έρευνας στο πλαίσιο αυτό. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές στα μέτρα που λαμβάνουμε και τα σχέδια που προχωρούμε. Στον ορίζοντα 2020 συμπεριλάβαμε τη συνέργεια με άλλα ταμεία, περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά ταμεία, να συγχωνευτούν και να συγκλίνουν οι προσπάθειες σε σχέση με τα κράτη-μέλη, ώστε να εξευρεθεί μια πρακτική μορφή ε, συνέχισης, ώστε να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός χώρος ερεύνας, όχι μόνο στα λόγια ή θεωρητικά ή φιλοσοφικά, αλλά ως αρχές στην πραγματική του εφαρμογή. Και το ίδιο, το πακέτο οι δέσμοι για την καινοτομία είναι πολύ σημαντική υπόθεση και μπορεί να συνεισφέρει και στο ε, πλαίσιο της πρόθεσης της έρευνας. Ε, η ιδιωτική και δημόσια συμμετοχή, η συνεργασία ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις ΔΙΤ και επίσης η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε σχέση με την έρευνα. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα και πρέπει να τύχουν συνέχεια. Και για το διάστημα Έχουμε και το ίδιο πρόβλημα σε σχέση με τον ορίζοντα 2020. Μεγάλη αύξηση από πλευρά κονδυλίων και στον ορίζοντα 2020 ένα νέο πρόγραμμα SSD το οποίο ακόμα δεν είναι απόλυτα σαφές από πού θα αντληθούν κονδύλια για να προχωρήσει αυτό. Κατά τους πρώτους μήνες λοιπόν της εφαρμογής όλων αυτών οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρετε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Η κυρία Μαντουρέλ παρακαλώ. Sí, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας. Προφανώς έχετε αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και σίγουρα επικροτώ το πρόγραμμά σας. Είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σαφείς στόχους αύξησης της ε, ανταγωνιστικότητας για την ευρωπαϊκή επιστήμη και την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και επικροτώ επίσης την πρόταση που έγινε για την τεχνική επιστημονική συνεργασία στη Μεσόγειο, μια φιλοδοξία που σκεφτόμασταν και αναπτύσσαμε εδώ και πολλά χρόνια και που πιστεύω ότι αποτελεί μια πολύ καλή ιδέα που θα είναι σημαντική για την ελληνική προεδρία, ό,τι και να συμβεί. Ε, η Πεσόγειος είναι μια σημαντική περιοχή της Ευρώπης. Η κυρία Καρβάλιο μίλησε για το πρόγραμμα Horizon 2020. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό ξανά. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με το πακέτο καινοτομίας και τα νομοθετικά πακέτα εταιρική σχέση που θα εγκρίνουμε αύριο το πρωί στην Επιτροπή, εν ώψη ιδίως των τριλόγων που θα ξεκινήσουν αμέσω μετά. Πρώτον, να σας πω κύριε Υπουργέ ότι παρότι οι κανονισμοί που επηρεάζουν τα PSP πρέπει να περάσουν με συναπόφαση, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι αποτελούν ένα ενιαίο πακέτο. Και με αυτή την προσέγγιση δουλέψαμε όλες οι πολιτικέ ομάδες στο Κοινοβούλιο. Η ομάδα μου το είπε και προηγουμένω στον Υπουργό Μεταφορών θεωρεί ότι οι εταιρικέ αυτέ σχέσει αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για το πρόγραμμα πλαίσιων ορίζοντας 2020, ιδίως δε διότι πετύχαμε αρκετές ε, συμφωνίες στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και προσπαθούμε τώρα να ενσωματώσουμε τις συμφωνίες αυτές στους κανονισμούς. Συμφωνίες που πραγματικά, κύριε Υπουργέ, είναι αποτέλεσμα, και το είπε και η κυρία Καρβάλιο, είναι αποτέλεσμα ε, σκληρής εντατικής δουλειάς πολλών μηνών. Και η εμπειρία που αποκτήσαμε θα είναι χρήσιμη νομίζω για τις εταιρικές σχέσεις πρώτης γενιάς και είμαστε πεπισμένοι ότι τα νέα κείμενα βελτιώνουν τα σημαντικά αυτά εργαλεία ως προς τη διαφάνεια και μια σειρά άλλων πραγμάτων που δεν θα αναφέρω τώρα. Ωστόσο, θέλουμε, θα θέλαμε, το Συμβούλιο να λάβει υπόψη, όπως το έκανε ήδη στις διαπραγματεύσεις για το Horizon 2020 κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας, το ζήτημα αυτό εμείς τις τοπολογίες μας αυτό που θέλαμε να περάσουμε ε, ιδίως για το στοιχείο των, της χρηματοδότησης, τα εργαλεία αυτά είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι λιγότερο σημαντικά τα ανταγωνιστικά συνεργατικά έργα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα σε κάθε challenge να υπάρχει κατανομή ισορροπημένη των διαφόρων ε, τομέων. Δεν μιλήσω παραπέρα. Ήθελα να κάνω και άλλη ερώτηση, αλλά μου με σταματάει η πρόεδρος, θα το αφήσω να το κάνουν οι συνάδελφοι. Ελπίζω κύριε Υπουργέ να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα που έχουμε ενώπιόν μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη, αλλά κοιτάω και το ρολόι που και που, οπότε δεν μπορώ να ε, αφήσουν να προχωρήσει ο χρόνο. Έχουμε και άλλε παρεμβάσει και μετά πρέπει να απαντήσει και ο υπουργό. Ο κύριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ περιορίζομαι όμω σε κάποιε παρατηρήσει SST. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει ο τρίλογος. Θα ήθελα να υπάρξει ειδική χρηματοδότηση. Δεν είναι πολύ μεγάλα κονδύλια. Πιστεύω ωστόσο ότι μαζί με την ε, δραστηριότητα εντοπισμού και δορυφόρων και υποδομών μπορούμε να ξεκινήσουμε και με μια θετική δράση από τροχιοποίηση των ε, δομών αυτών, διότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε τόσο πολύ εντατικά στο διάστημα που πρέπει να είμαστε όσο πιο ασφαλείς γίνεται από πιθανούς κινδύνους συγκρούσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης πολύ σημαντικό είναι όλα όσα είπατε για τα PPP και τις κοινοπραξίες και τις ε, κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές ως ε, λίκνα διαμόρφωσης προηγμένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Και εδώ νομίζω το έχετε τονίσει κι εσείς. Πολλά άλλα θέματα υπάρχουν. Όλο το ζήτημα, για παράδειγμα, του τριλόγου σήμερα το απόγευμα και κατά πόσον θα υπάρξουν ε, βήματα μπρος στο SST. Η κυρία Χέτζοκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Υπουργέ, εδώ βρίσκομαι. Έχετε δύσκολο έργο ενώπιον σας, επειδή καθώς ήμουν εισηγήτρια, συντάκτρια γνωμοδότησης για το κεφάλαιο 1α για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, κανένας πιθανότατα δεν ξέρει καλύτερα από μένα ότι έχουμε έλλειψη κονδυλίων εκεί και δεν είμαστε έντιμοι περί αυτού. Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει ποιον μπορούμε να κρατήσουμε και ποιον θα αποπέμψουμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να είσαστε στεναρός, να μην εν, ε, ενδώσετε. Τον 21ο αιώνα χρειάζεται μια πολιτική για το διάστημα η Ευρώπη. Μην υπαναχωρήσετε. Το να βρεθεί ένας κακός συμβιβασμός δεν είναι καλή λύση. Να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλιστούν τα κονδύλια. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε τμήμα του χρονορίζοντα 2020. Όταν χρειάζονται ε, φρέσκα χρήματα, νοπά χρήματα, πρέπει από μια ενδιάμεση αναθεώρηση να προέλθουν. Μην ενδώστε και το εγκαταλείψετε. Αν εγκαταλείψουμε την έρευνα θα εγκαταλείψουμε τα πάντα. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά που έχουμε. Υπάρχει έλλειψη κονδυλίων θα πρέπει να δούμε σε σχέση με τον συμβιβασμό. Να μην ενδώσουμε, να μην εγκαταλείψουμε την αρχική μας απόφαση επί της αρχής. Θέλω ένα πράγμα να αναφέρω. Η διεύρυνση της συμμετοχής ε, κυρίως θα πρέπει να ισχύει για τα νέα κράτη-μέλη που δεν έχουν άλλο τμήμα του χρονορίζων 2020 για να συμμετάσχουν. Παρά αυτό, αν τους αντλήσουμε, τους πάρουμε αυτά τα χρήματα από αυτούς, τότε να είσαστε σίγουροι ότι στο Συμβούλιο θα έχετε μείζον πρόβλημα. Τα, οι υπουργοί των νέων κρατών μελών ε, θα ε, ε, είναι λοιπόν θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Ο συμβιβασμός ο οποίος ελήφθη ήταν κακός. Αλλά δεν μπορεί να επιληθεί με το να παίρνουμε χρήματα εμβαλωματικά από εδώ ή από εκεί, μικρά κονδύλια για να καλύψουμε ανάγκες. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η έρευνα στην Ευρώπη και πρέπει να διασφαλίσετε αυτή την έρευνα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Τελευταία. κύριε Χίμπνερ. Ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε. Πρόκειται για την ανάπτυξη, την έρευνα, την καινοτομία, θέματα που είναι της αρμοδιότητας. Σας θέλω εδώ να αναφερθώ στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Όμως το 2013 θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει ένα ξεχωριστό έγγραφο για κάθε ερευνητικό Ινστιτούτο. Πώς θα οργανωθεί η συνεργασία με τις χώρες που είναι πιο παλιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτές που προσχώρησαν πιο πρόσφατα. Και κάτι άλλο τώρα. Με ποιο τρόπο και που σκοπεύετε να υποφεληθείτε από το πρόγραμμα ανταλλαγών έρασμος και την ανταλλαγή των ασκούμενων. Ο θεσμός της άσκησης επιτρέπει στους νέους να αποκτήσουν εμπειρία και είναι ένα σημαντικό εργαλείο, γιατί εκεί παίρνουν μαθήματα για ολόκληρη τη ζωή τους, που τους είναι χρήσιμα σε ολόκληρη τη ζωή τους. Οπότε πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα. Πολλές ερωτήσεις, λίγος χρόνος ε, κύριε Υπουργέ. Θα ζητήσω από τους γερμηνείς να μας δώσουν λίγο περισσότερο χρόνο και σας δίνω το λόγο. Ε, ε, πρέπει να σας πω ότι επειδή είστε υπουργός, ε, είστε και υπουργός θρησκευμάτων. Εγώ καθολική είμαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι έσχατοι έσονται πρώτοι αναγκαστικά. Κύριε Υπουργέ. Η κυρία Καρβάλιο πράγματι έθεσε με έναν τρόπο σωστό και τις, ε, καταρχήν την, ε, την ευθυγράμμιση που έχουμε και έτσι πρέπει να είναι σε πολλά από τα ζητήματα που αφορούν αυτόν τον κρίσιμο τομέα αλλά βέβαια και το γεγονός ότι έχουμε ε, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και ιδιαίτερα τις νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε ένα διάστημα το οποίο είναι και συντμημένο γιατί ερχόμαστε σε μια Προεδρία που έρχεται με το τέλος αυτού του Κοινοβουλίου και άρα οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Και εδώ ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει προεργασία και γίνεται ε, πολύ εντατική προσπάθεια και νομίζω ότι με την συνδρομή όλων των ε, εμπλεκομένων θα μπορέσουμε να φέρουμε αυτές τις, την υλοποίηση όλων των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο εφήγει αφορά το ζήτημα της διαφάνειας, της συμπερίληψης α, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλα αυτά όμως τα οποία είναι πράγματι αποτελούν μέρος της πολιτικής βούλησης, γιατί και η εφαρμογή του προγράμματος α, εμπεριέχει ανοιχτή και πρόσκληση προς ανοιχτή πρόσκληση προς επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει και ε, πρόνοια και για την συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βέβαια αυτό το οποίο αναφέρατε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή η απλούστευση των κανόνων ή των, και των διαδικασιών. Και επίσης η, ορίζοντας ε, θα χρηματοδοτήσει και συνεργατικά βέβαια χρησιμοποιώντας και πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, για να ολοκληρώσω την απάντηση, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε πλήρη επίγνωση του περιορισμένου χρόνου αλλά και του έμπρος των νομοθετικών πρωτοβουλειών θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθούν και ήδη είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο σε όλα τα σημεία και υπάρχει και σύγκληση απόψεων σε πάρα πολλά πράγματα. κυρία Μαντουρέλ, ε, βεβαίως το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη ε, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν ε, ακόμη πολύ προσοχή αυτό το οποίο, αυτά τα οποία είπατε και βέβαια πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία όσον αφορά την κατανομή και των τομέων. Συμφωνώ απολύτως. Όσον αφορά το θέμα της του Space Surveillance Tracking, το οποίο έθεσε ο, ο κύριος Πρόντι. Πράγματι, είναι προφανές ότι με τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει από την Ευρώπη, σε προγράμματα όπως το Κοπέρνικους και τον Καλίλαιο, αυτά γίνονται πλέον ιδιοκτησία, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως όλες οι ιδιοκτησίες, όλες οι υποδομές χρειάζονται ένα tracking, χρειάζονται έναν έλεγχο, χρειάζεται, χρειάζονται μια ασφάλιση, <laughs> μια προσοχή, μια ασφάλεια, μια προσοχή. Άρα αυτή είναι μια μείζον επιλογή θα έλεγα η προστασία των ε, υποδομών μας και γι' αυτό ο, ο νομοθετικός φάκελος ο SST είναι μια από τις προτεραιότητες ε, για μας. Βασιζόμαστε στη συνεργασία με τα ε, με τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Αναφερθήκατε στην χρηματοδότηση και βλέπουμε ότι υπάρχουν βέβαια μεγάλες διαφορές χρηματοδότηση, αν δούμε τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ξοδεύουν τεράστια ποσά όσον αφορά το ανάλογο πρόγραμμα και είναι φυσιολογικό, έχουν ε, πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και πολύ πιο μακρόχρονη αν θέλετε επένδυση. σε εμά πράγματι τα ε, κονδύλια αυτά θα πρέπει σιγά σιγά να αυξηθούν γιατί αποτελεί πλέον ε, μια σημαντική πολιτική της Ένωσης. Η κυρία Χέρτσοκ ε, έκανε ε, νομίζω σημαντικά, σημαντικές επισημάνσεις όσον αφορά το θέμα, της, όσον αφορά το θέμα των χρηματοδοτήσεων, όσον αφορά το θέμα των περικοπών του προϋπολογισμού και πώς αυτό θα επηρεάσει και ποιους και τα οποία ακούμε με μεγάλη προσοχή και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη γιατί ε, πράγματι η, πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία είναι ίσως από τις πλέον σημαντικές πολιτικές της Ευρώπης, αφορά όλους και βέβαια εμείς μας, πάντοτε μας ενδιαφέρει η διεύρυνση της συμμετοχής. Τώρα, όσον αφορά α, τις παρατηρήσεις της κυρίας Χίμπνερ, το, η συνεργασία ε, με τον, ε, με τον ιδιωτικό τομέα νομίζω ότι και αυτή είναι μια σημαντική πολιτική έρχεται να δώσει αν θέλετε και τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας και ανάπτυξη είναι μια, είναι μια πρωτοβουλία είναι οι, άτυπες, οι, οι συμπράξεις αυτές είναι πολύ σημαντικές και ε, αυτό το οποίο αναφέρεται όσον αφορά το ζήτημα της συμμετοχής και όσον αφορά το θέμα της μεταχείρισης, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει, ακούμε με προσοχή, συζητάμε, για να βρούμε μια, μια βέλτιστη λύση. Αλλά πάντως όλα αυτά όπως έχουν γίνει μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, έτσι και συνεχίζονται στο διάλογο μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής αλλά ε, και του Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να έχουμε και με τα συμπεράσματα τα οποία ε, έχετε υιοθετήσει και την ψηφοφορία που θα γίνεται να έχουμε πάντοτε την ε, χρυσή τομή, δηλαδή την οδό αυτή η οποία θα είναι προώθηση των κοινών μας στόχων. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη γιατί σας πιέσαμε χρονικά. Πρέπει να πω ότι και η συνάντηση αυτή που εκτιμούμε ιδιαίτερα μαζί σας όπως και με τους προηγούμενους συναδέλφους μαρτυρεί την δέσμευση της ελληνικής προεδρίας ε, την παρουσία της οποίας εκτιμήσαμε ήδη και στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να ξέρετε ότι θα, έχετε από πλευράς μας στενή συνεργασία τους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς που μείναν περισσότερο. Θυμίζω ότι θα συνεχίσουμε το απόγευμα στην αίθουσα, στο κτίριο Γιάν, όπως ε, σας είπα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Grazie. Grazie. Gli που purtroppo. <laughs>